Dear colleagues, let us start. Αγαπητοί συνάδελφοι, ας ξεκινήσουμε την απογευματινή μας συνεδρίαση. Λοιπόν, με ποια σειρά θα εξετάσουμε τώρα τις αναφορές. Έχει υπάρξει μια αλλαγή ακούσουμε πρώτα την 367 του 2018, Αριάννα Καλανέλα, για το δικαίωμα εργασίας ανθρώπων με αναπηρία. Η αναφέρουσα δεν είναι παρούσα, επομένως θα δώσω κατευθείαν το λόγο στην εκπρόσωπο της Επιτροπής, με Πλαθένσια Κορέρο είναι η εκπρόσωπο τη ε, Επιτροπή. Παρακαλώ, έχετε το λόγο κυρία Πρωθυπουργέ Κορέρο. Σύντομα, πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η κατάσταση είναι δύσκολη και υπάρχει ένα, ε, ε, μια δυσκολία στην εξέβρεση εργασίας των ανθρώπων με αναπηρία προσπαθεί να αξιοποιήσει τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της για να βελτιώσει την κατάσταση αυτή. Προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να ενημερώσουμε για την οδηγία η οποία προστατεύει τα άτομα με αναπηρία μεταξύ άλλων από, την, ε, από τις διακρίσεις στον χώρο εργασίας και εξειδικεύουμε την έννοια ε, των εύλογων ρυθμίσεων για τα άτομα με αναπηρία. Συλλέγουμε επίσης στατιστικά στοιχεία και όσον αφορά ε, τα, τις αναπηρίες, αλλά επίσης ε, όσον αφορά το φύλλο και την ηλικία. Να αναφερθώ επίσης και στον πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Σύμφωνα με την αρχή 17, αναγνωρίζεται το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να ε, έχουν ένα περιβάλλον εργασίας προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους. Ε, θα ήταν ευχή έργο να μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε και απευθεία με την αναφέρουσα, αλλά αυτό έχουμε να δηλώσουμε μέχρι στιγμή. Σα ευχαριστούμε. Υπάρχουν ήδη συνάδελφοι που έχουν ζητήσει το λόγο και θα ξεκινήσουμε από τον κύριο Ντούντα. Γιάροσλαφ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, κύριε και κύριοι, στην Ευρώπη έχουμε πάνω από, ένα, 100 ε, εκατομμύρια άτομα με αναπηρία και αυξάνεται αυτός ο αριθμός. Χρειάζεται λοιπόν να βρούμε τρόπου έτσι ώστε όλα αυτά τα άτομα με αναπηρία να μπορούν να συμμετέχουν στην οικονομική, κοινωνική ζωή, να βρίσκουν δουλειά και να μπορούν να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο αυτόνομα. Είναι απολύτω απαραίτητο να το καταφέρει αυτό η Ευρώπη. Δεν είναι απλώ μια υποχρέωση που έχουμε αναλάβει επειδή επικυρώσαμε το σύμφωνο του για τα δικαιώματα ατόμων με αναπηρία, αλλά επίση γιατί αποτελούν αυτοί οι άνθρωποι και ένα δυναμικό κοινωνικό, οικονομικό, πνευματικό για την Ευρώπη. Η υποχρέωση των ευλόγων ρυθμίσεων στο περιβάλλον εργασίας σημαίνει ότι θα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στα άτομα με αναπηρία να εκφράζουν τις δικές τους δεξιότητες, να αποκτούν νέες δεξιότητες, και να τους δώσουμε όλα τα εφόδια που χρειάζονται για να μπορέσουν να συμμετάσχουν στην αγορά εργασίας. Η συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας είναι ο καλύτερος τρόπος να ε, προλάβουμε το ενδεχόμενο να περιπθωριοποιηθούν κοινωνικά και οικονομικά. Γι' αυτό ζητώ να κρατήσουμε την αναφορά ανοιχτή, τουλάχιστον μέχρι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημοσιοποιήσει το προσχέδιο της στρατηγικής της για τα άτομα με αναπηρία μετά το 2021. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε. να Γκέμα, επόμενη μιλήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Αριάννα, ε, δηλαδή η κοπέλα η οποία υπέβαλε την αναφορά, είναι πολύ σημαντική, πολύ σοβαρή ε, και ε, αυτή τη βδομάδα στην ε, ε, στο γραφείο μου ήρθε ένα, ένα νέο παιδί, ο Εμμανουέλε, ο οποίος ε, είχε ε, προβλήματα ε, ιδιαίτερα και από τότε που ήταν φοιτητή μέχρι και τώρα, όπως ο Εμμανουέλ ή η Αριάννα, πολλά είναι τα παιδιά με αναπηρίες τα οποία αρρωσταίνουν ακριβώς λόγω της ανεργίας και εν τέλει γίνονται πρόβλημα για την κοινωνία που τα αντιμετωπίζει τα παιδιά αυτά σαν αντικείμενα χωρίς να τους ε, δίνει ε, δυνατότητα προσωπικής ε, και εργασιακής πρόθεσης. Η πρόσβαση λοιπόν στην αγορά εργασίας για άτομα με αναπηρία εξακολουθεί να είναι προβληματική με πάρα πολύ ψηλό ποσοστό πολύ ψηλό ποσοστό ε, σε σχέση με τα άτομα που δεν έχουν αναπηρία. Ε, επομένως, ε, δεν μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να ζήσουν μια ζωή ανεξάρτητη. Θα πρέπει οπωσδήποτε να ενεργήσουμε με τρόπο ώστε η Σύμβαση των Ανθρωπίνων των Ηνωμένων Εθνών για τα άτομα με αναπηρία να ε, εφαρμόζονται σε όλες τις χώρες και μάλιστα με τον ίδιο τρόπο έτσι ώστε να μην υπάρξει καμία και να μην υπάρχει καμία διακριτική μεταχείριση. Θα πρέπει να σταματήσει οποιαδήποτε διάκριση ε, όσον αφορά τα εργασίες εργασιακές δυνατότητες, να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες, ε, δικαιώματα όσον αφορά τα ε, συνδικάτα ε, και επαγγελματική κατάρτιση. Ζητώ να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά βάσει και της εργασίας που έχει ξεκινήσει για την στρατηγική για την αναπηρία μετά το 2020. Τα, και θέλουμε τα άτομα με αναπηρία να έχουν εν να επιτύχουν εν τέλει αυτήν την πρόσβαση στην αγορά εργασίας που επιθυμεί η αναφέρουσα. Ευχαριστώ πολύ. Ε, έχουμε πολλούς καταγεγραμμένους, εγγεγραμμένους μάλλον ομιλητές, ο κύριος Μάριο Φουρών. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εγώ αποφάσισα να μιλήσω ε, υπέρ αυτής ε, της ε, αναφοράς καθότι τα θέματα αυτά περί αναπηρίας αφορούν εμάς όλα τα θεσμικά όργανα και κυρίως την Επιτροπή μας. Η Αριάννα Κολονέλο, έχουσα ειδικέ ικανότητες, καταγγέλει αυτή τη στιγμή την σύμβαση που τους αναγνωρίζει ίδια δικαιώματα όσον αφορά την απασχόληση και που έχει παραμείνει κενό γράμμα. Εξακολουθούν να παραμένουν αποκλεισμένοι από την αγορά εργασία στα περισσότερα κράτη-μέλη. Επομένως, η νομική ε, αρχή της ισότητας μπορεί να υπάρχει, αλλά στην ουσία ε, ε, πραγματικά δεν μπορεί να συμβάλλει η ίδια στη βελτίωση της κοινότητας και της κοινωνίας. ο, ο χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων το, της Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκής Ένωσης βασίζεται ε, στην αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης και της σταθερότητας. Εντός του 2020 προβλέπει η νέα στρατηγική ότι θα πρέπει να ε, ξεπεραστούν τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν άτομα με αναπηρία. Ζητούμε για όλους αυτούς τους λόγους να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά. Ο κύριος Ακούς ε, Σαλίμπα. Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, το δικαίωμα στην εργασία δεν είναι καπρίτσιο. Αποτελεί ε, αρχή οικονομικής και κοινωνικής ανεξαρτησίας. Το να είναι κανείς αποκλεισμένος λόγω της αναπηρίας του αποτελεί διακριτική μεταχείριση για τα εργασιακά, σχετικά με τα εργασιακά δικαιώματα. Υπάρχει άρρωστη, άλλωστε η σχετική ε, συνθήκη την οποία εμείς έχουμε προσυπογράψει ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, επομένως, ε, και ως κράτη-μέλη που έχουν ε, υπογράψει την συνθήκη, γιατί και μεμονωμένα έχουν υπογράψει αυτή τη συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών, ε, είμαστε υποχρεωμένοι και δυνάμει του άρθρου 27 να δίνουμε τις ίδιες ευκαιρίες στα άτομα με αναπηρία. Θα πρέπει λοιπόν με σαφή και ρητό τρόπο να πούμε ότι όλοι οι άνθρωποι με αναπηρία ή όχι θα έχουν ε, ισότιμη πρόσβαση ε, στην εργασία. Η ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών επιθυμεί η αναφορά αυτή να παραμείνει ανοιχτή και ε, προβλήματα όπως αυτά τα οποία αναφέρονται σε τούτη ε, την αναφορά να ρυθμιστούν στην στρατηγική για την αναπηρία που θα καλύψει την περίοδο 2020 με 2030. Θα πρέπει να σταλεί ένα ισχυρό μήνυμα στο σύνολο των κρατών μελών έτσι ώστε ε, να ρυθμιστεί σε επίπεδο κρατών μελών και Ευρωπαϊκής Ένωση, αυτό το πρόβλημα της διακριτικής μεταχείρισης. Η προσβασιμότητα είναι πάρα πολύ σημαντική ε, και η έλλειψη ε, υποστήριξης αυτών των αναπήρων είναι πολύ σοβαρό πράγμα. Πρέπει οπωσδήποτε να τους βοηθήσουμε να ενταχθούν στην κοινωνία. Πρέπει με τρόπο ολοκληρωμένο να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Να μείνει παρακαλώ ανοιχτή αυτή η αναφορά. Köszönöm szépen a lehetőséget, Είμαι πάντα ευτυχής ε, όταν μιλάμε για αναφορές με τέτοιο περιεχόμενο. Συμφωνώ απολύτως ε, και με αυτά που είπαν οι προλαλήσαντες συνάδελφοι. Δεν θέλω να τα επαναλάβω. Δεν θέλω να επαναλάβω και την βασική αρχή ε, που είναι ακριβώς η σύμβαση για, την, για το δικαίωμα στην εργασία. Εγώ μελέτησα την αναφορά και η αναφέρουσα ε, είναι νομικός, ε, πολύ καλά καταρτισμένη, ε, αλλά δυστυχώς από τη στιγμή που έχει προβλήματα όρασης δεν μπορεί να βρει δουλειά. Και αυτό που έχω να πω είναι ότι υπάρχει πρόβλημα εδώ, ε, γιατί δεν υπάρχει άλλωστε και ομοιομορφία μεταξύ των κρατών μελών. Δεν υπάρχουν ελάχιστες προϋποθέσεις. Ε, σήμερα το πρωί μιλήσαμε για τα εκλογικά δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία και νομίζω ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε την ίδια πορεία, δηλαδή να καθοριστούν και για τις υπηρεσίες και για, τις, ε, την αγορά εργασίας και τα εργασιακά δικαιώματα ελάχιστα στα ε, δικαιώματα τα οποία θα είναι εναρμονισμένα. Ελπίζω ότι μετά από 10 χρόνια στρατηγικής για τους αναπήρους ε, αυτή ε, η στρατηγική θα περιλάβει ακριβώς τέτοιες διατάξεις ε, που θα οδηγήσουν σε εναρμονισμένη αντιμετώπιση. Ευχαριστώ πολύ και θέλω να μείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά έτσι ώστε να την αντιμετωπίσουμε με μεγαλύτερη σοβαρότητα και ενδελεχώς. Ευχαριστώ. Thank you, Ευχαριστούμε κύριε Κώστα. Θα ήθελα και εγώ να μιλήσω εκ μέρου και τη ομάδα των Πρασίνων. Υποστηρίζουμε και εμεί την πρόταση να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά. Δεν θα συμφωνήσω με το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε η εκπρόσωπο τη Επιτροπή. Δεν μπορείτε να αυτοεξαιρίστε αν θέλετε από τη δημιουργία ενός μηχανισμού παρακολούθησης του τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Βεβαίως υπάρχει ένας ανεξάρτητος μηχανισμός στο πλαίσιο του ΟΗΕ που θα παρακολουθεί τις δεσμεύσεις που ανελήφθησαν στο πλαίσιο της σύμβασης του ΟΗΕ. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέτασε αυτό αυτή τη σύμβαση του ΟΗΕ. Έχουμε και συγκεκριμένο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την, που, το, την υποστηρίζει. Και υπενθυμίζω λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι έχει και εκείνη υποχρέωση να παρακολουθήσει την εφαρμογή α, α, αυτών των διατάξεων, αυτού, με ένα μηχανισμό τον οποίο να τον... Ε, ε, ο οποίο να αξιοποιεί μάλλον όλα τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση συμπεριλαμβανομένων και του Κοινοβουλίου. Μήπω οι εκπρόσωπε τη Επιτροπή θα ήθελαν να κάνει κάποιε επιπλέον παρατηρήσει, μια και δεν είναι εδώ λοιπόν η αναφέρουσα. Ερχόμαστε στο συμπέρασμα. Η πρόταση είναι να παραμείνει η αναφορά ανοιχτή. Επίση, προτείνεται να αποσταλούν ε, επιστολέ στο Συμβούλιο και στι εθνικέ αντιπροσωπείε, υπενθυμίζοντα και ζητώντα του στοιχεία για τι ε, ρυθμίσει που πρέπει να και τα μέτρα που θα πρέπει να αναλάβουν για τη διευκόλυνση της ε, επασχόληση των ατόμων με αναπηρία. Επίσης, θα να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθήσει σε ποιο βαθμό τα κράτη-μέλη έχουν ενσωματώσει στο εθνικό τους δίκαιο τη σχετική οδηγία και να επανέλθει στο μέλλον με περισσότερες πληροφορίες, δεδομένου ότι προτείνουμε να παραμείνει η αναφορά ανοιχτή. Δεν άκουσα κάποια διαφορετική πρόταση, επομένως θα λέω ότι μάλλον συμφωνούμε, έτσι να παραμείνει ανοιχτή και θα αποστείλουμε και τις επιστολές που ανέφερα. Και με την ευκαιρία της παρουσίας της, των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα τους επιθυμίσουμε και τις δικές τους αρμοδιότητες σε σχέση με την παρακολούθηση τέτοιων δεσμεύσεων. Σας ευχαριστώ. περάσουμε στην επόμενη, που ήταν το προηγούμενο σημείο της ημερές διάταξης. ή από την Ισπανία για τη Βαλένσια και τους καλλιεργητές πορτοκαλιών. Είναι 280 του 2019. Ο κύριος Λουκ Μπερλετιέ από την Κομισιόν. Euh, Ευχαριστώ πολύ. Ναι, γνωρίζουμε πολύ καλά την σημασία που έχει ε, ο τομέα των σπεριδοειδών στην Ισπανία γενικότερα και στην Βαλένθια ειδικότερα. Επανειλημμένα και πέρσι και φέτο ενημερωθήκαμε για την κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί σε αυτήν την ε, περιοχή. Μάλιστα συναντήσαμε εδώ στις Βρυξέλλες και τους παραγωγούς. η ε, παραγωγοί της περιοχής της Βαλένθια αναφέρονται σε προβλήματα όσον αφορά τα εσπυροδοειδή της περιοχής τα οποία ε, εικάζουν ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω των εισαγωγών από τη Νότια Αφρική. Ε, οι στατιστικέ όμω που έχουμε στη διάθεσή μα δείχνουν ότι μακροοικονομικά δεν έχει υπάρξει αύξηση τη εισαγωγή εσπεριδοειδών από τη Νότια Αφρική προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιθέτως υπάρχει μείωση. Στο έτος 2018 είναι γεγονό ότι είχαμε κατά 5% αυξημένε εισαγωγέ από την περίοδο Οκτώβριο νοεμβριο που είναι η περίοδος παραγωγής εις την Βαλένθια. Αντιθέτως όμως εκείνη την περίοδο ε, ε, μειώθηκαν ε, πάρα πολύ και αν πάρουμε την, τους, τα στοιχεία για το 19 οι εισαγωγές από την Νότια Αφρική είναι κατά 10% μειωμένες σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Εάν υπάρχει λοιπόν ένα πρόβλημα στο στα Ισπυριδοειδή στην Ισπανία σαφώ δεν οφείλεται στι αγωγέ από τη Νότια Αφρική. Αντιθέτως, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι υπήρξαν προβλήματα διαρθρωτικά στην περιοχή παραγωγής της Βαλένθια. Το 18-19 η παραγωγή ε, ήταν πολύ μεγάλη στην περιοχή αυτή. Είχαμε σοδιές κατά 8% αυξημένες σε σχέση με την προηγούμενη εσοδεία. Υπήρξαν επίσης κλιματολογικές συνθήκες ε, οι οποίες οδήγησαν σε καθυστέρηση στην ορίμανση των ε, σπυριδοειδών και επομένως είχαμε σε μικρότερη χρονική περίοδο περισσότερο προϊόν που έπρεπε να πουληθεί. Επίσης ε, ε, η ποιότητα ήταν πιο χαμηλή γιατί είχαμε μικρότερου μεγέθους περιδοειδοί. Υπήρξαν επίσης ε, ε, λόγω κλιματικών συνθήκων ε, μικρότερη ζήτηση ε, γιατί είχαμε ένα χειμώνα λίγο πιο ήπιο, πιο ζεστό. Τέλος, υπήρξαν ισχυρές βροχοπτώσεις καθώς επίσης και πλημμύρες που προκάλεσαν φυτοϊγειονομικά προβλήματα και επομένως οδήγησαν σε αρκετά χαμηλό ή εν πάση περιπτώσει χαμηλότερο από το συνηθισμένο ε, ε, επίπεδο ποιότητας. Ε, όλα αυτά δημιούργησαν προβλήματα όσον αφορά την εμπορία εσπεριδοειδών από την Ισπανία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, όταν συναντήσαμε τους παραγωγούς της Βαλένθια εδώ στις Βρυξέλλες, σημειώσαμε ότι υπάρχει και ένα πρόβλημα οργάνωσης του τομέα ε, της ε, εσπεριδοπαραγωγής ε, στην Βαλένθια. Το ποσοστό οργάνωσης των παραγωγών φτάνει στο 34%, χαμηλό λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν στην Ισπανία 300 περίπου, 300 περίπου οργανώσεις παραγωγών που ε, υποστηρίζονται κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και που ε, μπορούν να επενδύσουν μέσω επιχειρησιακών προγραμμάτων. Εάν οι επαγγελματίες δεν οργανώνονται σε οργανώσεις παραγωγών, δεν έχουν πρόσβαση ε, σε, αυτά τα, σε αυτούς τους πόρους και επομένως δεν μπορούν επίσης να αντιμετωπίσουν λύσουν προβλήματα φυτοϊγειονομικά μέσω συγκεκριμένων βοηθημάτων, μέσω μέτρων κρίσης κλπ. Υπάρχουν επίσης ε, ε, προγράμματα ανάπτυξης της υπαίθρου, καθώς επίσης και κάποια προγράμματα επένδυσης ε, που καλύπτονται από το γενικότερο προγραμματισμό ανάπτυξης της υπαίθρου. Επομένως, αυτοί που βρίσκονται εγκατεστημένοι στην περιοχή της Βαλένθια έχουν στη διάθεσή τους εργαλεία και μέτρα τα οποία θα τους δίνουν την δυνατότητα να διαχειρίζονται κρίσεις, κυρίως δε κρίσεις παραγωγής, ε, καθώς επίσης και να βελτιώνουν τον, την ανταγωνιστικότητά τους μέσα από επενδύσεις ε, περιβαλλοντικού χαρακτήρα ή επενδύσεις ε, που αφορούν τα φυτογειονομικά, καθώς επίσης και τι υποδομές. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την, την επεξήγηση. Δεν ξέρω ποιος θέλει να πάρει το λόγο. Κυρία Ρέκο. Ευχαριστώ. Είναι σίγουρο ότι αυτή η επιστολή, αυτή η αναφορά που μας έστειλαν οι παραγωγοί της Βαλένθια είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα που μας δείχνει πώς αυτές οι συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου επηρεάζουν την καθημερινότητα των μικρών παραγωγών στην Ευρώπη και εν προκειμένου στην Ισπανία. Εγώ με, με από τις εξηγήσει που μας έδωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής. Γιατί, Κανείς, γιατί δεν αναφέρθηκε καθόλου στις συνθήκες υπό τις οποίες παράγονται τα εσπεριδοειδή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί στην Ένωση ζητάμε από τους αγρότες μας να κάνουν ιδιαίτερες προσπάθειες ε, και ξέρετε ότι το ζήτημα αυτό μας ανησυχεί και συζητείται ευρέως στις χώρες μας. Εξάλλου, μια, ένα από τα αιτήματα των συνδικαλιστικών οργανώσεων των παραγωγών είναι ακριβώς αυτό. Και είναι σημαντικό να το φέρουμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχει η, η ρήτρα ε, στην συμφωνία που υπογράψαμε με το, το 2016 με την Νότια Αφρική ρήτρα για τον τρόπο με τον οποίο θα ελέγχεται η διαδικα... η... ο αντίκτυπος που μπορεί να έχει αυτή η εμπορική συμφωνία και ότι θα υπάρχει ένα, ένας μηχανισμός με διαφάνεια, ότι θα διευκολύνεται η ετικετοθεσία, ότι θα είναι ξεκάθαρα το φύτιο υγειονομικό καθεστώς και, το, και επίσης ότι θα είναι ξεκάθαρη η προέλευση του προϊόντος. Δηλαδή έχουμε εργαλεία στη διάθεσή μας για να επιλύσουμε τα προβλήματα που θέτει ο αναφέρον. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν εμείς ζητούμε να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά και να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια έκθεση που να μας εξηγεί πώς και γιατί δεν έχει εφαρμοστεί αυτή η ρήτρα ε, ε, ασφαλείας, safety clause, στην συμφωνία με την Νότια Αφρική του 2016. Γιατί δυστυχώς αυτή τη στιγμή οι παραγωγές περιοδών της Βαλένθια αναγκάζονται να αντιμετωπίσουν έναν αθέμητο ανταγωνισμό. Ευχαριστούμε. Επόμενη μιλήτρια η κυρία Γκυλιάρ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όπως αναφέρει ο αναφέρον, η κατάσταση της παραγωγής περιδοειδών στη Βαλένθια είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Έχουν να αντιμετωπίσουν η παραγωγή μια κατάσταση όπου τους, που τους έχει οδηγήσει να πουλούν κάτω του κόστους ε, εδώ και χρόνια έχουν να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό όχι μόνο από την Νότια Αφρική αλλά και από την Αίγυπτο εξαιτία των συμφωνιών ελευθέρου εμπορίου και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει αντιμετωπίσει αυτόν τον ανταγωνισμό αποτελεσματικά. Αυτό θέτει σε κίνδυνο το μέλλον αυτών των ανθρώπων, αυτών των παραγωγών. Ακούμε καθησυχαστικά μηνύματα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωστόσο, ε, δεν είναι συμπληρωματικές αυτές οι αγορές σε πολλές περιπτώσεις, να σας δώσω ένα παράδειγμα, τον Αύγουστο άρχισαν να εμφανίζονται πορτοκάλια που ερχόντουσαν από άλλες χώρες, από τρίτες χώρες. Εμείς όμως το φθινόπωρο, τελευταίο γίνεται η σοδιά. Ε, Επίσης υπάρχουν μεγάλες διαφορετικές διαφορές στη, στα ημερομίσθια. 10 με 12 είναι ε, ευρώ τι, τι, είναι το ημερομίσθιο των εργατών στη Βαλένθια, ενώ είναι υποπολαπλάσιο στις χώρες όπως στη Νότια Αφρική ή άλλες. 50 σεντ την ώρα. έχουν λοιπόν να αντιμετωπίσουν αυτόν τον αθέμητο ανταγωνισμό που φτάνει στα επίπεδα τη μια μαύρη αγορά. Και τι μα απαντά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε ήδη τα πρώτα ε, δείγματα μειώνονται το εισόδημά τους, ότι ε, ε, έχουν να αντιμετωπίσουν ε, προβλήματα φυτοϊγειονομικά, όπως για παράδειγμα το πρόβλημα με τη μεριλανική λίδα. Θα ήθελα λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, να ζητήσουμε να παραμείνει η αναφορά ανοιχτή και να ζητήσουμε περισσότερες πληροφορίες από την Επιτροπή. Γκαρθία Μαργάγιο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Τα σπυριδοειδεία αντιμετωπίζουν μεγάλα προγράμματα. Εγώ θα αναφερθώ μονάχα σε δύο. Ε, η μερολόγιο, ας πούμε, εσοδείας παραγωγής ε, και συμφωνίες. Μέχρι πρόσφατα η μοναδική ε, το που μας απασχολούσε στην Βαλένθια ήταν η Τουρκία και το Μαρόκο, Βόρεια Αφρική κλπ. Ενώ εδώ και μερικά χρόνια έχουμε και επίσης τα, τις εισαγωγές από την Νότια Αφρική. Πρώτον έχουμε ε, την ε, παραγωγή ε, μανταρινιού που ήταν μηδενική τότε όταν υπεγράφει η συμφωνία και έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Δεύτερον, γιατί έχει εν, ε, ε, έχει διευρυνθεί η περίοδος εισαγωγής μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, πράγμα που επικαλύπτει, ε, την δικιά, τη δικιά μας παραγωγή. και μάλιστα έχουμε εισαγωγές με διευκολύνσεις τελωνιακές. Τα στοιχεία εσωτερικής παραγωγής, καθώς επίσης και ο, η εισαγωγή των μανταρινιών και των πορτοκαλιών είναι ένα μεγάλο ε, πρώτο πρόβλημα και αναφέρεται στην αναφορά. Το δεύτερο είναι το πρόβλημα των ε, των ασθενειών. Ε, δεν είναι καλός ο έλεγχος των εσπεριδοειδών από την Νότια Αφρική. Είναι ελληματικό ο έλεγχο και ήδη έχουν βρεθεί ε, διάφορες ε, ε, νόσοι φυτογενομικού χαρακτήρα και επομένω αυτό μας προβληματίζει το πρώτο στοιχείο, το πρώτο μέρος της ε, αναφοράς ήδη είναι προβληματικό. Το δεύτερο ε, είναι ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να, ε, οι κοινοτικοί οργανισμοί να προχωρήσουν σε ελέγχους φυτοϊγειονομικούς. Κοιτάξτε, εμείς ε, η Υποδέμωση, η Vox και εμείς του ΕΛΚ μιλάμε ε, με, το, με τα ίδια λόγια και πρέπει να σας πω ότι αυτό είναι ένα θαύμα, δεν έχει γίνει ποτέ και ακόμα και αυτό το γεγονός από μόνο του θα πρέπει να σας οδηγήσει στα συμπεράσματα που ε, πρέπει. Ευχαριστώ πολύ. Mr. Ah, Ο κύριος Βάσκης Λάθαρα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. 125.000 ε, παραγωγή και χιλιάδες εκτάρια. Ε, ε, η Ισπανία είναι η πρώτη χώρα παραγωγός φρέσκων πορτοκαλιών, μανταρινιών και άλλων εσπεριδοειδών. Αυτό αποτελεί πλούτο όχι μονάχα για την Ισπανία αλλά και για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να υποστηριχτεί από αυτήν. Γι' αυτό λοιπόν συμφωνούμε ε, και μοιραζόμαστε τον προβληματισμό του τομέα που δυναμητίζει την ευζοία του τομέα αλλά και όσων ασχολούνται με αυτόν. Οι εισαγωγές από την Νότια Αφρική ε, έχουν επιδεινώσει την κατάσταση, ωστόσο δεν είναι η μοναδική αιτία ε, και γι' αυτό δεν θα πρέπει να περιοριστούμε σε αυτό ως αιτία του προβλήματος. Ξεκινάμε στους επόμενους μήνες τις διαπραγματεύσεις για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Εμείς ζητάμε μια κοινή γεωργική πολιτική η οποία ε, θα υποστηρίζει τους παραγωγούς που θέλουν να εξυγχρονίσουν ε, τις ε, εκμεταλλεύσεις τους και να δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία. Θα πρέπει να βασιστούμε στην ποιότητα και όχι μονάχα στις χαμηλές τιμές. Στις μελλοντικέ οικονομικές συμφωνίες με την Μεγάλη Βρετανία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την ε, μεγάλη, το μεγάλο ποσοστό εξαγωγών στην χώρα αυτή. Και αυτό θα πρέπει να ληφθεί οπωσδήποτε υπόψη. Τέλος, θέλουμε να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να ε, ενεργοποιήσει τις ρήτρες para compensar a τις ρήτρες ε, ασφαλείας ε, και σε περίπτωση που αυτές οι ρήτρες δεν γίνονται σεβαστές κυρίως όσον αφορά τον έλεγχο υγειονομικό και φωτογειονομικό να ενεργοποιήσει τις, ε, τα απαραίτητα μέτρα. κοιτάξτε, εμείς δεν θεωρούμε το ελεύθερο εμπόριο ως κάτι απαραίτητα αρνητικό αλλά οπωσδήποτε δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι θα πρέπει να δώσουμε όλες τις δυνατότητες ε, στην Ισπανική Γεωργία. Ευχαριστώ. Next, Mr. Ben Κύριος Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Προσυπογράφω απόλυτα όσα είπαν οι προηγούμενοι Ισπανοί συνάδελφοι. Η παραγωγή μπήκε σε ένα τομέα και επειδή μειώνονται, ε, το, μειώνεται το εμπόριο από τις άλλες χώρες, δεν σημαίνει ότι βελτιώθηκε η κατάσταση. Δηλαδή μπορεί κατά 10% να αλλάξει η τιμή, αν αλλάξει κατά 1% το εμπόριο, μειωθεί ε, ή αυξηθεί. Ε, όπως είπαμε, πρέπει να προσέχουμε το ύψος του κόστους παραγωγής σε ορισμένες χώρες και η παραγωγή στην Ισπανία είναι ακριβότερη. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι η παραγωγή είναι υπό ίδιες συνθήκες. Και επίσης, ε, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για την προστασία των φυτών, τα ευρωπαϊκά προϊόντα, η ντόπια παραγωγή στην Ευρώπη ε, ε έχει ε, καλύτερο καθεστώς, καλύτερη θέση από τις εισαγωγές από άλλες χώρες. Και αυτό ενδιαφέρει πολύ την υγεία. Όπως είπε και η Κομισιόν, υπάρχουν διάφορες δυνατότητες ούτως ώστε οι οργανώσεις παραγωγών και η εμπορία να ενισχυθούν ε, και μέσα από αγροτικούς ε, συνεταιρισμούς ε, μεταξύ άλλων. Εγώ θα ήθελα να πω για την ομάδα μου ότι κρατάμε ανοιχτή την αναφορά και περιμένουμε από την Κομισιόν να μας υποβάλει πλήρη έκθεση. Ευχαριστώ. Η κυρία Γιέρα Καρσία. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνούμε λοιπόν όλοι συνάδελφοι. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω όμως και για ένα ζήτημα στο οποίο αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στα εσπεριδοειδή διαπιστώνουμε ότι η παραγωγή είναι μικρότερη από τη ζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή στην Ευρώπη δεν παράγουμε όσα εσπεριδοειδή ε, χρειαζόμαστε, θέλουμε να, θέλουμε να καταναλώνουμε. Ωστόσο, υπάρχουν λοιπόν για αυτό το λόγο εισαγωγές από τρίτες χώρες. Και ιδιαίτερα εδώ μιλούμε για την Νότια Αφρική η οποία έχει άμεσες επιπτώσεις στο, στην παραγωγή, στους παραγωγούς σπυριδοειδών στην Ισπανία και αλλού. Βεβαίως μπορεί να υπάρχουν δομικά προβλήματα σε αυτό το τομέα όπως και σε άλλους. Όμως, οι τελευταίες συμφωνίες οδήγησαν σε σημαντικές αλλαγές και αυτό θα πρέπει να το αναγνωρίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εάν όχι η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου, τουλάχιστον η Γενική Διεύθυνση Αγροτική Ανάπτυξη. Θα πρέπει κάπω να το εκτιμήσει. Ε, φτάνουμε ε, μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Δηλαδή, μια περίοδο ε, στην οποία υπάρχει αλληλεπικάλυψη των εισαγωγών με την περίοδο που υπάρχει παραγωγή στη Βαλένθια. Και το λέω αυτό και στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπήρξαν δύο περιστατικά την προηγούμενη χρονιά που μειώθηκαν οι οι δασμοί για τα εσπεριδοειδή τα οποία εισάγονται για τη χρήση, αυτών των, για τη χρήση των εσπυροειδοειδών από τη μεταποιητική βιομηχανία. Και γιατί συμβαίνει αυτό. Και γιατί συμβαίνει αυτό ιδιαίτερα με μια χώρα όπως η Νότια Αφρική, η οποία έχει μια ιδιαίτερα επικίνδυνη προϊστορία με το, τα φυτογειονομικά, όπου έχουμε μια ασθένεια επικίνδυνα, την, τη μελανική λίδωση, και η οποία μπορεί να έχει επιπτώσεις. Τόσο μεγάλες που μπορεί να οδηγήσουν στο να χαθεί μια ολόκληρη σουδιά. Γιατί. Συμβαίνουν όλα αυτά γιατί υπάρχουν συμφέροντα τα οποία επιθυμούν να προωθήσουν τις εισαγωγές από την Νότια Αφρική. Ο, ο, στόχος θα έπρεπε να είναι να ε, ε, ζητήσουμε, να απαιτήσουμε από την Νότια Αφρική να βελτιώσει τις συνθήκες παραγωγής. Και αυτό ε, πρέπει να το αναγνωρίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι ένα αίτημα του κλάδου των παραγωγών της Βαλένθια. Υπάρχουν λοιπόν αυτά τα δύο προβλήματα. Αυτή η αύξηση του χρόνου του ε, παραγωγής με αποτέλεσμα να υπάρχει επικάλυψη με την ε, περίοδο παραγωγής στη Βαλέφια και τα προβλήματα που αφορούν στις εισαγωγές. Και ταυτόχρονα λοιπόν έχουμε μειώσει τους δασμούς για εισαγόμενα από την Νότια Αφρική. Αυτό είναι λοιπόν κίνδυνο, είναι πρόβλημα για την ευρωπαϊκή παραγωγή, βεβαίω και είναι. Αυτού του τύπου τα προβλήματα δημιουργούνται με τέτοιου τύπου συμφωνίες. Όχι μόνο, δεν είναι μόνο σε σχέση με την Νότια Αφρική, αλλά στην, περίπτωση των εσπυριδοειδών είναι ιδιαίτερα ε, με την Νότια Αφρική γιατί αν δεν αναλάβουμε δράση, τι θα πετύχουμε, τι, τι σκοπεύουμε να κάνουμε, να καταστραφεί τελικά όλη η παραγωγή στην Ευρώπη. Υπάρχουν λοιπόν οι επιπτώσει αυτών των συμφωνιών στον ευρωπαϊκό και πιο συγκεκριμένα στο, στον, στην παραγω, στους παραγωγούς της Βαλένθια. Όπως λοιπόν και όλοι οι συνάδελφοι, βλέπετε υπάρχει πλειοψηφία, ζητούμε και εμείς να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά και υπενθυμίζω στην Ολομέλεια είχαμε εγκρίνει ένα ψήφισμα με το οποίο δεν, έδωσα, δεν, δεν εγκρίναμε ε, την, ε, δεν εγκρίναμε την πράξη κατεξουσιοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα επέτρεπε σε ε, εσπεριδοειδή από την Νότια Αφρική με χαμηλότερα πρότυπα φυτογενομικά να εισάγονται. Γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια σύγκρουση ανάμεσα στα συμφέροντα των παραγωγών, του κλάδου της παραγωγής αυτού της Νότιας Αφρικής και των συμφερόντων των Ευρωπαίων παραγωγών. Δεν υπάρχουν άλλοι ομιλητές. Κλείνουμε λοιπόν. Όλοι ε, ζητούν να μείνει ανοιχτή αναφορά για τις ε, σχετικές επιτροπές αυτή η αναφορά πήγε στην Άγκρη στις 20 Νοεμβρίου και στην Ίντα επίσης στις 20 Νοεμβρίου. Η Άγκρη δεν απάντησε. Η Ίντα απάντησε και είπε ότι η Ίντα αποφάσισε την αναφορά να τη λάβει υπόψη στο συνεχιζόμενο έργο της Επιτροπής. Υπάρχει και γραπτή απάντηση της Κομισιόν, αλλά μας τα είπε και ο εκπρόσωπος της Κομισιόν. Ε, από 18 Φεβρουαρίου είναι η απάντηση και λέει η Κομισιόν, η Κομισιόν ε, δεν πιστεύει ότι είναι δύσκολη η αγορά υπήρχε, ότι αυξήθηκε δηλαδή η εισαγωγή από από τη Νότια Αφρική. Υπάρχει δηλαδή μια αμφισβήτηση εδώ μεταξύ των δύο θέσεων. Οπότε αυτό από μόνο του συνιστά λόγο για να δοθεί συνέχεια στο θέμα ώστε να πάρουμε πιο πολλές πληροφορίες. Άρα η ε, αναφορά παραμένει ανοιχτή και δεν ξέρω να ξαναστείλουμε, να ξαναστείλουμε την επιστολή στην Άγκρη ίσως υπενθυμίζοντάς τους ότι δεν έχουν ακόμη απαντήσει, εντάξει. Εκτός μικροφώνου παρέμβαση. Εσείς είστε μέλος της Άγκρη, οπότε εσείς ίσως πρέπει να επιμείνετε. Ναι, εγώ είμαι μέλος, όμως όπως και ένα σωρό άλλοι συνάδελφοι. Όλοι εμείς είμαστε μέλη της ε, Επιτροπής. Εγώ, εγώ, ναι, εγώ οπωσδήποτε και χωρίς αμφιβολία ε, θα ε, κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου. Θα ήθελα την ίδια προσπάθεια να καταβάλει και η ομάδα των Πρασίνων, παρακαλώ. Ωραία θα κάνετε επαφή όλοι με την Άγκρη ως μέλη αυτής της Επιτροπής και θα δώσετε συνέχεια. Πάμε παρακάτω τώρα εμείς. Τι έχουμε. Ε, αναφορά 886-1168 του 2016 και η 1059 του 2019. Διάφοροι Ισπανοί πολίτες διατήρηση του Μαρμενόρ. Οι αναφέροντες, οι δύο αναφέροντες είναι εδώ. η κυρία Ιζαμπέλ Ρούμπιο Περές. Για πέντε λεπτά maximum. Εγώ δεν είμαι Ιζαμπέλ Ρούμπιο, αλλά είμαι δικηγόρος της... Α, μάλιστα, εσείς ε, αντιπροσωπ... αντιπροσωπεύετε, εκπρόσωπος νομικός. Ευχαριστώ πολύ. Η περιοχή της Μούρθια, όπως και πολλές άλλες περιοχές, βλέπουν αυτήν την εκατόμβη, ε, μία ε, αυτοκτονία οικολογική, η οποία ε, οδηγεί σε μεγάλα προβλήματα τις, τις, τους κατοίκους της περιοχής. Όταν στα τέλη του, 17, του 16 υποβάλαμε αυτήν την αναφορά, το Ιμάρ Μενόρ είχε έναν υπερβολικό ευτροφισμό. Ε, μετά από πολλές διαπραγματεύσεις ε, σε αυτήν την Επιτροπή ε, είδαμε ότι υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη έλλειψη ισορροπίας του οικοσυστήματος. Επίσης, επανειλημμένα στην περιοχή είχαμε πλημμύρες λόγω των υπογείων υδάτων ε, καθώς επίσης και λόγω των προβλημάτων οικοδόμησης ε, και της ανάπτυξης που η ρίστο εμπαρόδο είναι, ε, είναι παράνομη. Οι Ισπανικές αρχές αλλά και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έδωσαν διάσταση ιδιαίτερη στο θέμα δηλώνοντας ότι όλα τα μέτρα διοικητικά και άλλα είχαν ληφθεί έτσι ώστε να μην ε, υπάρξει αυτή η οικοκτονία ε, όπως την ονομάζουμε εμείς η περιφέρεια της ε, ε, Μούρθια έκανε ε, μαζί με αντίστοιχους οργανισμούς μετά από καταγγελίες των κατοίκων ανέλα, έκανε, πήρε κάποια μέτρα ωστόσο δεν ελήφθησαν πραγματικά υπόψη τα όσα είχε αρχικά πει η υδρογραφική υπηρεσία της Σεγούρα. Ε, επίσης δεν ελήφθησαν μέτρα ε, σχετικά με την ε, νητρορύπανση. Αυτή τη ε, στιγμή έχουμε 9.600 εκτάρια τα οποία έχουν αναγνωριστεί ως παράνομα από την υδρογραφική ε, Υπηρεσία της ε, Σεγκούρα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη και κατεπίγουσα. Λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι τα προληπτικά μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος δεν έχουν ληφθεί υπόψη καθότι οι αρμόδιες αρχές σε για θέματα νητρορύπανση δεν έχουν λάβει τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα, ούτε και τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα, ε, ε, θεωρούμε ότι υπάρχει παραβίαση των, ε, του, του νομοθετικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όσον αφορά την προστασία των περιοχών Natura 2000 και όσον αφορά επίσης την, τις οδηγίες για τα ύδατα. Αυτή τη στιγμή σε αυτήν την ε, περιοχή που είναι μία από τις ε, ε, πιο... Es una etiqueta formal que no responde a una gestión eficiente de lo que sería una zona de... που είναι μία από τις πιο άνυδρες περιοχές, έχουν αναπτυχθεί εκτάσεις εντατικής καλλιέργειας αυτή τη στιγμή παραβιάζεται ακόμα το άρθρο 6 της, ε, ε της οδηγίας ε, Habitats, καθώς επίσης ε, και της οδηγίας για τα πτηνά. και επομένως δημιουργούνται ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. η περιβαλλοντική ζημία της, του Μαρ Μενόρ ή ως αποτέλεσμα της ρήπανσης λόγω των λιμάτων τα οποία φθάνουν και συσσωρεύονται λόγω των υδατορευμάτων είναι πάρα πολύ μεγάλη μεγάλη. Τέλος, διαπιστώνουμε ότι εδώ και χρόνια ε, δεν λαμβάνονται υπόψη είναι ε, και ε, τα ευρωπαϊκά περιβαλλοντικά μέτρα, δημιουργώντας μεγάλο πρόβλημα και στο οικοσύστημα, αλλά και όσον αφορά την υγεία των ατόμων. Ε, εδώ βρισκόμαστε ε, στο, ε, στον οίκο της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας έτσι ώστε να ακουστεί η φωνή μας. Θέλουμε να καταγγείλουμε την διοικητική ανοχή η οποία δολοφονεί την Μαρ Μενόρ καθώς επίσης και το γεγονός ότι οι αρμόδιες αρχές δεν επαγρυπνούν ως οφείλουν. Εδώ χάνουμε ένα οικοσύστημα το οποίο γνωρίζουμε από την παιδική μας ηλικία ε, και το οποίο προσπαθούμε να προστατέψουμε γιατί είναι η δικιά μας Μαρμενόρ. Τέλος, ε, ε, λόγω της ε, ιδιαίτερα επικίνδυνης κατάστασης θεωρούμε ότι θα πρέπει να διασφαλιστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα τα οποία συνδέονται με την ζωή της Μαρμενόρ και του περιβάλλοντος. Η δικιά, το δικό μας αίτημα είναι να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά. Θα πρέπει επίσης να υπάρξουν συστάσεις έτσι ώστε να αντιστραφεί η καταστροφική πορεία ιστορία ε, του Μαρμενόρ ε, και θα θέλαμε να ασχοληθεί με το θέμα και η Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίση, ζητούμε από την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει μια διαδικασία επιπαραβάση ειδικά για τη Μαρμενόρ. Χρειάζεται ενεργητική παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε να μπορέσουμε να σώσουμε ένα μοναδικό ε, ε, σύστημα, οικοσύστημα ε, στο, το, στο οποίο ζουν χιλιάδες άνθρωποι. Ευχαριστώ. Είναι πρόσφατη αυτή η αναφορά του κυρίου του, έχουμε, του 19 Λούις Αλβαρές. Δεν βλέπω τον αναφέροντα να είναι εδώ. Είναι εδώ. Για πέντε λεπτά, όχι περισσότερο. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας που μας δίνει τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε αυτή την αναφορά για την κατάσταση στη Μαρμενόρ. Μια αναφορά που ελπίζουμε να τύχει προσοχής. και ελπίζουμε να μας βοηθήσετε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση της πλήρους, του, να έχει αγνοωθεί πλήρως αυτή η περιοχή εδώ και 30 χρόνια από όλα τα θεσμικά όργανα. Μια εγκατάλειψη η οποία συνεχίζεται και η οποία δυστυχώς συνεχίζεται ε, και ελπίζουμε να μην συνεχιστεί. Το πρώτο πρόβλημα είναι το γεγονό ότι η Ισπανία δεν σέβεται τι δεσμεύσει τη σε σχέση με μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος. Τα μέτρα που προβλέπονται στο, στη στρατηγική της διαχείρισης των υδάτων λέγεται από τις παρεμφυριακές αρχές ότι λύνουν το πρόβλημα. Ωστόσο, αν δείτε το άρθρο 4 του οδηγίας πλαίσιο για τα υδατά, περιγράφονται τα όρια που θα πρέπει να τηρούνται για την ε, κατάσταση των υδάτων και πράγματι οι περιφερειακές αρχές έχουν ε, αναλάβει μια σειρά μέτρων τεχνικών και νομικών για την αντιμετώπιση της ε, μόλυνσης στη Μαρμενόρ. Πρώτα απ' όλα δημιουργήθηκε μια επιστημονική επιτροπή. Υπήρξε επίσης ένα διάταγμα για την προστασία της Μαρμενόρ που υιοθέτησε μια σειρά υποχρεωτικών μέτρων για την γεωργία στην περιοχή ειδικά για την περιοχή του Μαρμενόρ. Ωστόσο, ελπίζουμε ότι η ουσιαστική εφαρμογή της ε, ε, Ευρωπαϊκής Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας θα οδηγήσει στην επίλυση των προβλημάτων του Μαρμενόρ. Αυτά μας λένε οι περιφερειακές αρχές, αλλά δεν είναι αλήθεια. Δεν έχει λειτουργήσει η Επιστημονική Επιτροπή, δεν έχουμε επιτροπή ε, με την οποία να συμμετέχουν οι πολίτες χρειάστηκαν χρόνια για να εγκριθούν τα σχέδια και οι στρατηγικές που επιβάλλεται να υπάρχουν με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Στοιχεία τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα για να θεωρηθεί ότι το κράτο εκπληρώνει τι υποχρεώσει του με βάση αυτέ τι ευρωπαϊκές οδηγίε. Δυστυχώ λοιπόν σήμερα βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη κατάσταση, η οποία έχει επιδεινωθεί τον προηγούμενο Σεπτέμβριο από τι πλημμύρε. Και καταδεικνύει αυτό ότι ότι το σχέδιο διαχείρισης της Μαρμερών δεν είναι αποτελεσματικό. Τα τελευταία δυόμισα χρόνια είχαμε ε, τρία νομοθετήματα για τη διαχείριση της γεωργίας στην περιοχή, που σας δείχνει πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση. Ο κάθε νόμος όμως τροποποιεί τον προηγούμενο. Το ζήτημα είναι να υπάρξει έλεγχος τη μόλυνση στην πηγή της και διαχείριση της αγροτικής και αστικής χρήσης της γης. Με μέτρα επιστημονικά τεκμηριωμένα. Αυτή τη στιγμή έχουμε μόλυνση από νητρικά. Και αυτή είναι η κυριότερος, ο κυριότερος λόγος της υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Και παρόλα αυτά δεν έχει αναλευθεί ούτε ένα μέτρο για την αντιμετώπιση της μόλυνσης από, το, τα λοιπάσματα, από τα νητρικά. ούτε η ε, ε, κυβέρνηση η εθνική έχει υπάρξει ε, πιο αποτελεσματική από την περιφερειακή. Αν δείτε το σχέδιο διαχείρισης των υδάτων, μόνο 7 από τους στόχους εκπληρώθηκαν και 10 ξεκι... Μάλλον, 17 από τα μέτρα από τα 100 μέτρα που περιλαμβάνει έχουν εκπληρωθεί, ενώ όλα αυτά θεωρούνταν απαραίτητα για την διαχείριση της ποιότητας των υδάτων στη Μαρμενόρ. Το 2016 είχαμε το νέο σχέδιο και είχαν ήδη παρατηρηθεί προβλήματα με τον ευτροφισμό ήδη από το καλοκαίρι του 2016. Αυτός ο ευτροφισμός έχει οδηγήσει στην ενεργοποίηση εσωτερικών μηχανισμών του οικοσυστήματος που έχει επιδεινώσει την κατάσταση. Θεωρούμε λοιπόν ότι συντρέχουν οι υποθέσεις του παραγράφου 4 του άρθρου 4 της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Διαχείριση των Υδάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρούμε ότι επίσης μπορεί να ε, θεωρηθεί ότι υπάρχει παραβίαση του, της έκτης παραγράφου του ιδίου άρθρου. Σας ζητούμε επίσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επισκεφθεί την περιοχή της Μούρθια. Να στείλει μια αποστολή ευρωβουλευτών για να αντιληφθείτε και μόνοι σας την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή αυτή. Θα δείτε ότι η φύση προσπαθεί να μας μιλήσει και δυστυχώς εμείς οι άνθρωποι δεν την αφουγκραζόμαστε. Ευχαριστώ. Εκπρόσωπος της Κομισιόν, ο κύριος Χωσέ Μαρία Ράμος Φλωρίντο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, τους ε, αναφέροντες ε, για την παρουσίασή τους. Η Κομισιόν πάντα ακούει όλες τις απόψεις. Αυτή τη στιγμή όμως είναι πολύ χρήσιμο που σας ακούμε έτσι ώστε να επικαιροποιηθούν οι πληροφορίες που έχουμε για την περίπτωση αυτή. Θα ήθελα να πω ότι βεβαίως η Κομισιόν γνωρίζει την μεγάλη οικολογική σημασία της Μαρ Μενόρ που έχει μεγάλη σημασία και σε ευρωπαϊκή ευρωπαϊκό επίπεδο και βεβαίως είναι εμβληματική σημασία για την περιοχή της Μούρθια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμερίζεται τον προβληματισμό για τις πιέσεις που υφίστανται η Μαρ Μενόρ ε, ε, και που οδήγησε σε ε, το οικοσύστημα σε ακραίες καταστάσεις και κατεπίγουσα εν πάση περιπτώσει κατάσταση. Το πρόβλημα έρχεται από παλιά, το είπαν και οι ομιλητές, το 2016 υπήρξε μια ιδιαίτερη κρίση χημική και οικολογική και από εκείνη τη στιγμή η Μενόρ αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα μεγάλης ε, σημασίας ε, όπου τον, ε, το φθινόπωρο του 19 επιστεγάστηκαν, ακορυφώθηκαν μάλλον με ιδιαίτερες βροχοπτώσεις και πολλές πλημμύρες. Ε, οπωσδήποτε η μεγάλη ε, δραστηριότητα, ανθρώπινη δραστηριότητα στην περιοχή αυτή έχει επιδεινώσει την κατάσταση. Αλλά από το 2016 ε, έχουν γίνει πολλές μελέτες, έχουν γίνει πολλές αναλύσεις. Η επιστημονική κοινότητα εξακολουθεί να αναλύει την κατάσταση. Έγκριτοι επιστήμονες, καθηγητές έκαναν μια διάγνωση της κατάστασης. Ε, και ε, πρόσφατα ελήφθησαν ε, σχετικά μέτρα από τις τοπικές περιφερειακές αρχές. Σε αυτά θα αναφερθώ αργότερα. Θα ήθελα ε, ε, όμως εγώ κυρίως να σας πω τι έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα τελευταία χρόνια σε σχέση με το θέμα. Πρώτα απ' όλα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κράτησε ανοιχτό διάλογο με τις Ισπανικές Αρχές όσον αφορά την κατάσταση της Μαρ Υπήρξαν συναντήσεις στις Βρυξέλλες με τις περιφερειακές αρχές καθώς επίσης και με τις εθνικές αρχές ε, στην Μαδρίτη και στην Μούρθια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστήριξε οικονομικά και επιστημονικά τις ε, εν λόγω αρχές ε, στην, αντιμετώπιση, στην προσπάθεια αντιμετώπισης του προβλήματος. Θέλω δε να πω ότι στα πλαίσια της ε, αρχής ε, της επιτήρησης ε, της εφαρμογής της, της οδηγίας έχουμε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υπενθυμίσει στις περιφερειακές αρχές ότι υπάρχουν η οδηγία για την φύση, η οδηγία για τα ύδατα και η οδηγία για την νητρορύπανση. Αυτές είναι οι τρεις οδηγίες που μας ενδιαφέρουν εδώ και σε Mm. Ε, ε, σε μία έκθεση την οποία ε, έδωσε στο Κοινοβούλιο, παρέδωσε στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρεται ιδιαιτέρως στην οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα και την εφαρμογή της και αναφέρεται στο, κεφάλαιο 6 συγκεκριμένα στην Ισπανία. Στον τρίτο κύκλο υδρογραφικής διαχείρισης για την περίοδο από το 2021 έως το 2027 ε, πιστεύουμε ότι θα ληφθούν ε, ιδιαίτερα μέτρα ε, όσον αφορά τη λεκάνη απορροής στη συγκεκριμένη περιοχή. Ε, επίσης, ε, ε, δεν μιλάμε μόνο για συστάσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άνοιξε και δύο διαδικασίες επί παραβάση εναντίον της Ισπανίας και μετά μεταξύ άλλων και στην Μούρθια και σε κοινότητες οι οποίες είναι σημαντικές για τη Μαρμενόρ. Μία διαδικασία σχετικά ε, με ελλειπή εφαρμογή της οδηγίας για την ε, νητρορύπανση. Δόθη παρά ε, περιθώριο αντίδρασης από την Ισπανία, καθότι αυτή δεν, η Ισπανία δεν ελέγχει σωστά τα ύδατά της και οπωσδήποτε όσον αφορά την νητρορύπανση θα πρέπει να ληφθούν επιπλέον μέτρα. Ως, διαδικασία, ως απόρρια της διαδικασίας αυτής επιπαραβάσει. Ε, με διάταγμα της 23 ε, Νοεμβρίου ε, στην Μούρθια ορίζονται νέες ευαίσθητες περιοχές όσον αφορά την νητρορύπανση, ε, ε, διευρύνονται οι φυστάμενες περιοχές ε, και λαμβάνεται υπόψη η παράκτια περιοχή της Μαρ Μενόρ ως ιδιαίτερα, περιοχή ιδιαίτερης νητρορύπανσης. Καταλαβαίνουμε βεβαίως ότι αυτό δεν είναι αρκετό, δηλαδή αφού οριστούν οι ευάλωτες ζώνες θα πρέπει οπωσδήποτε να υλοποιηθούν ε, μέτρα κατάλληλα έτσι ώστε να μειωθεί η νητρορύπανση. Η διαδικασία επιπαραβάση έχει ξεκινήσει και συνεχίζει την ε, πορεία της και περιμένει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την συγκεκριμένη απάντηση από τις αρχές της Μούρθια. Δεύτερη ε, διαδικασία επιπαραβάση σχετίζεται με τις οδηγίες για τα οικοσυστήματα Habitat. Ξεκίνησε το 2015 καθότι ε, περιοχές ε, της ε, Natura 2000 ορίζονται ως περιοχές ιδιαίτερης συντήρησης και επομένως απαιτούν συγκεκριμένο πρόγραμμα διαχείρισης αυτών των ε, περιφερειών. Ε, μετά από πολλά σκαμπανεβάσματα, όπως είπα και προηγουμένως, τον Οκτώβριο του 2019 ενέκρινε ε, το σχέδιο ιδιαίτερων περιοχών συντήρησης η περιφέρεια της Μούρθια, συμπεριλαμβάνονται δε και περιοχές της Μούρθια και του Μαρμενόρ και αναφέρονται επίσης συγκεκριμένα μέτρα της παράκτειας μεσογειακής ζώνης της Μούρθια και κάποιες άλλες περιοχές. Ε, ε, ε, πρέπει να έρθουμε σε επαφή με τις Ισπανικές Αρχές για να δούμε εάν στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας που παραβάζει έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα. Επίσης, το Νοέμβριο του 2019 οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συναντήθηκαν στην Μαδρίτη με αρμόδιες εθνικές και περιφερειακές αρχές στα πλαίσια του σχεδίου δράσης για, την, για το περιβάλλον, την φύση, τους ανθρώπους και την εικόνα και αυτό ήταν απόρριο του fitness check των σχετικών οδηγιών που ανέφερα προηγουμένως. Αναφέρθηκε βεβαίως και η περίπτωση Μαρμενόρ και τα μέτρα συντήρησης, μαζί με άλλα πολλά ζητήματα. Οι Ισπανικές αρμόδιες αρχές δεσμεύτηκαν να στείλουν επιπλέον πληροφορίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά το θέμα αυτό, ωστόσο δεν έχουμε λάβει τίποτα προς ώρας. Εκτός από το νομικό ε, ζήτημα ε, και τις διαδικασίες επί παραβάση τις οποίες προσπάθησα να σας αναλύσω, πρέπει να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, μέσω κοινοτικής χρηματοδότησης προτίθεται να συμβάλλει στην ανανέωση, στην αναβίωση της ΜΑΡ Μενόρ. Αυτή τη στιγμή βέβαια το πιο σημαντικό είναι η, συμβολή των διαχρονικών ταμείων και των ταμείων συνοχής μέσω του ή τι ε, έτσι όπως ονομάζεται για τη Μάρα ε, Μενόρ. Ε, ήτι συμβαίνει ένα πρόγραμμα βάσει του οποίου διαφορετικά ευρωπαϊκά ταμεία δρούν για μια συγκεκριμένη περιοχή έτσι ώστε να υπάρξει οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη αυτής της περιοχές. Η Ισπανία έχει πολλές ΗΤΙΣ, μεταξύ των οποίων αυτή για την Μαρ Μενόρ και μέσω των μέτρων αυτών ε, ε, ε, στόχος είναι να ξεπεραστούν τα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα και να αναβιώσει οικολογικά η Μαρ Μενόρ. Επίσης υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι από τα διορθωτικά ταμεία, από το Ταμείο της Αλίας, το Ταμείο για την Ανάπτυξη της Υπέθρου, σε ύψος 70 εκατομμυρίων που μπορούν να μοχλεύσουν πολύ περισσότερα, ε, πολλούς περισσότερους πόρους. Ε, θα πρέπει βέβαια να δοθούν τα χρήματα αυτά με την προϋπόθεση ότι οι περιφερειακές και εθνικές αρχές της ε, Ισπανίας χρησιμοποιούν τα χρήματα αυτά, τους πόρους αυτούς για συγκεκριμένη μέτρα που θα οδηγήσουν στην αναβίωση της περιοχής. Ε, έχουν ληφθεί ήδη κάποια μέτρα τους τελευταίους μήνες από τις αρμόδιες αρχές ε, και επομένως δεν αναφέρονται, δεν συμπεριλαμβάνονται στην ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ας πούμε, ε, μέσω διατάγματος της 26ης Νοεμβρίου του 2019 η περιοχή της Μούρθια προωθεί ένα σχέδιο ολοκληρωμένης διαχείρισης της περιφέρειας της Μούρθια. Ε, και ε, αποφασίστηκε να περάσει για να εγκριθεί από το Κοινοβούλιο έτσι ώστε να γίνει νόμος που θα αρχίσει να ισχύει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης ε, αναλύει το περιεχόμενο αυτό, ε, αυτού του νέου νόμου για την προστασία της Μαρ Μενόρ. Ε, επίσης υπάρχει και το πρόγραμμα που λέγεται Πρόγραμμα Μηδενικών Λιμάτων για την Μαρ Μενόρ, για περιβαλλοντικό σχέδιο, το οποίο καθορίζει οδικό χάρτη με ένα ευρύ φάσμα μέτρων δίνοντας βεβαίως προτεραιότητα στα μέτρα αυτά τα οποία θα πρέπει κατά προτεραιότητα να ληφθούν έτσι ώστε να αντιστραφεί η κατάσταση. Επίσης πρέπει να σας πούμε ότι η εισαγγελία περιβάλλοντος της ε, Ισπανίας που ασχολείται με ιδιαίτερα σοβαρές καταστάσεις έχει ε, λάβει γνώση του θέματος ε, και έχει πολλές καταγγελίες που σχετίζονται με, το, με την ρήπανση της Μαρμενόρου. Μετά από όλα αυτά και εν συμπεράσματι, θα ήθελα να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να μελετά το θέμα πάντα εντός των πλαισίων των αρμοδιοτήτων της ε, και προσπαθεί να συμπεριληφθεί στην ε, ε, λύση του προβλήματος. Η ουσιαστική εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς επίσης και των μέτρων που απορρέουν από τις συγκεκριμένες περιβαλλοντικές οδηγίες είναι γεγονός ότι πρέπει να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την ιδιαίτερα περίπλοκη και κρίσιμη κατάσταση που αντιμετωπίζει ή Μαρ Μενόρ. Πάντα επί τη βάση των επιστημονικών ε, τεκμηρίων ε, πρέπει να ληφθούν οι σωστές ε, προτάσεις και μέτρα. Επίσης, Πρέπει να υπάρξει οπωσδήποτε αγαστή συνεργασία μεταξύ των ε, διαφόρων επιπέδων ε, ε, εκπροσώπησης τοπικού, περιφερειακού, εθνικού επίπεδου, καθώς επίσης και οπωσδήποτε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε πρόσωπε της Κομισιόν, Ράμος Φιωρίντο, ο λόγος στα μέλη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δυστυχώς, για άλλη μια φορά, συζητούμε αυτή την κατάσταση η οποία έχει χρονίσει. Θα ήθελα να συγχαρώ τους αναφέροντας και την πλατφόρμα τους, ε, την πρωτοβουλία τους, γιατί αν δεν υπήρχαν αυτές οι πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών, θα είχε παραμείνει άγνωστη η κατάσταση στο Μάρμελορ. Ευτυχώς λοιπόν υπάρχει η κοινωνία των πολιτών στις ε, επιτόπου, στα χωριά εκεί που προσπαθούν εδώ και χρόνια να αναλάβουν πρωτοβουλίε να λυθεί το πρόβλημα ενώ εμείς ακόμα το συζητάμε δυστυχώ. Και πράγματι πρέπει να το δει κανεί τι συμβαίνει για να το πιστέψει. Εγώ έρχομαι από τη Γρανάδα, βρίσκεται κοντά στη Μούρφια και πάνε ήδη 4-5 χρόνια όταν ξεκίνησε αυτή η κατάσταση, το 2016 όπως ακούσαμε, και ήταν τόσο σοβαρή που πραγματικά ε, είναι, είναι λυπηρό. Είναι πανέμορφης φυσικής ομορφιάς αυτή η λιμνοθάλασσα. Τότε λοιπόν, Αύγουστος του 2016, ακυρώθηκαν όλες οι κρατήσεις από τους τουρίστες, και ο κόσμος απελπίστηκε. Έτσι έχουν τα πράγματα. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται από τη μια στιγμή στην άλλη. δεν ξέρω πόσα προστατευτικά έργα και μέτρα υπήρχαν για την Λιμνοθάλασσα που είναι προφανές ότι δεν λειτουργήσαν. Και εγώ θα ήθελα να επισημάνω και το εξή. Α μην δείχνουμε ω υπεύθυνου και ένοχου του γεωργού, γιατί είναι και αυτοί που επλήγησαν. Όλοι οι γεωργοί έκαναν τα πράγματα σύμφωνα με τον νόμο. Τους έδινε άδειες η περιοχή, η αυτόνομη κυβέρνηση της Μούρθια για τις, τα αρδευτικά έργα, για όλες τις δραστηριότητες τους εκεί. Επομένως αυτό σημαίνει ότι είναι μια κατάσταση παρα... λανθασμένων επιλογών που κρατάει χρόνια. Εάν Επίσης, αν δεν τους είχαν δοθεί αυτές οι άδειε, δεν θα είχαν ακολουθηθεί αυτό το μοντέλο αγροτικής περιοχής στον κάμπο αυτόν. Τους οδηγήσαμε σε αυτήν την κατάσταση και ε, όλα, όλα, τους ε, ε γινόνταν γιατί επιτρέπονταν. Εγώ τότε ήμουν σύμβολος ε, κοινοτική στην σε, κοινότητα όμορη και θεωρούσαμε, το βλέπαμε ήδη ότι ο τρόπος με τον οποίο αναπτυσσόταν η περιοχή της Καρταχένα ήταν, δεν θα ήταν βιώσιμος. Πέρασαν χρόνια και ήλπιζα ότι θα αναλυθούν πρωτοβουλίε σε εθνικό επίπεδο για να επιληθεί η κατάσταση. Ζητώ συγγνώμη που μακρηγορώ. Ωστόσο, είναι προφανές ότι πρέπει να ληφθούν σοβαρά μέτρα. Ακούστηκε αυτή η πρόταση για να ξεκινήσει τη δικασία επί παραβάση όμως η κατάσταση έχει επίσης από την κλιματική αλλαγή. Ήδη αναφέρθηκε πριν από λίγους μήνες υπήρξαν τραγικές ε, φυσικές καταστροφές στην περιοχή της Καρταχένα. Υπάρχουν άνθρωποι που έμειναν άστιγοι από τις πλημμύρες. Και φυσικά όλα αυτά τα επηρεάζει και τα επιδεινώνει η κλιματική αλλαγή, αλλά πρέπει να κινητοποιηθούμε. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πιέσει γιατί όλα πρέπει να, πρέπει να αλλάξουν στην περιοχή. Και το μοντέλο της αγροτικής ανάπτυξης, αλλά και το μοντέλο της αστικής ανάπτυξης και επίσης το μοντέλο της τουριστικής ανάπτυξης σε αυτή την περιοχή. Γιατί όλοι αυτοί οι τομείς της οικονομίας έχουν συνεισφέρει με το πόσο με την απληστία, με την αρπακτικότητα με την οποία έχουν ε, καταστρέψει τους φυσικούς πόρους, στο να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Πριν από τέσσερα χρόνια εγώ δάκρυσα βλέποντας την κατάσταση στο Μαρ Μενόρ και ακούγοντας τους ανθρώπους εκεί να μου διηγούνται τι πέρασαν. Αλλά πριν τρία χρόνια, πριν δύο χρόνια συνέχιζαν να ε, δέχομαι ε, αιτήματα από τους συναδέλφους από τη ήρθε, έλα να δεις τι συμβαίνει, έλα να δει πώς συνεχίζεται η κατάσταση. Συνεχίζουμε να έχουμε ψαράδες που δεν μπορούν να ψαρέψουν η κατάσταση έχει φτάσει σε τέτοιο τραγικό σημείο που δεν είμαι σίγουρη αν μπορούμε να την αναστρέψουμε. Ελπίζω να είναι αναστρέψιμη, αλλά ελπίζω επίσης να λογοδοτήσουν, να δώσουν εξηγήσει όλοι αυτοί οι υπεύθυνοι, αρμόδιοι που φταίνε για αυτή την κατάσταση επί σειρά ετών. Γιατί είναι μια καταστροφή οικονομική, περιβαλλοντική ε, και κοινωνική άνευ ε, πιστεύω ότι θα μείνει στην ιστορία, στα, στα συγγράμματα για το πώς δεν πρέπει να αναπτύσσεται μια περιοχή, η περιοχή της Καρταχένα. Θα πρέπει να βάλουμε ένα ε, τέλος σε αυτή την κατάσταση. Βεβαίω υπάρχουν συνθήκε που έχουν διευκολύνει και επιδεινώσει την κατάσταση, αλλά θα πρέπει να κινητοποιηθούμε. πρέπει να κινητοποιηθεί η κυβέρνηση τη Ισπανία για να, για να επιλύσει αυτή την κατάσταση. Δεν ξέρω, σα το είπα, αν είναι αναστρέψιμη, αλλά εμείς από την πλευρά μας θα πρέπει να συνεχίσουμε να βοηθούμε αυτή την κοινωνία των πολιτών που ευτυχώ που την έχουμε για να μας ευαισθητοποιήσει, για να μας ξυπνήσει για την κατάσταση στο Μαρμενόρ. Ευχαριστώ. Μαρτίνε Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ο Μπαουθάντιας. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αναφέροντες που ήρθαν εδώ για να μας πούν την άποψή τους σε σχέση με την κατάσταση που αντιμετωπίζει τώρα η Μαρμενόρο και το πώς μπορούμε ε, να ε, την βελτιώσουμε. Θέλουμε ε, να σας καλωσορίσουμε γιατί εδώ είναι το σπίτι σας. Ε, και ε, είναι καλό που ε, και εμείς προσπαθούμε από τη δικιά μας τη μεριά και ανεξάρτητα από τον πολιτικό χώρο από τον οποίο προερχόμαστε να αντιμετωπίσουμε σαν Ισπανία το η Μαρ Ναι, βεβαίως βρίσκεται στην περιφέρεια της Μούρθια, ωστόσο η αποτελεί κληρονομιά όλων των Ισπανών και πρώτη η Μέρη Μουροθάλασσα μοναδική σε όλη την εγώ είμαι από τη Μαγιόρκα δεν είμαι από την Μουρθία, όλα αυτά έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα. Ακούγοντας ε, αυτά που ε, άκουσα, ε, πρέπει να σας πω ότι συμφωνώ με κάποια από αυτά που λέτε, γιατί και εγώ προσωπικά πριν από περίπου έξι μήνες ήρθα σε επαφή με μέλη της επιστημονικής κοινότητας και μάλιστα να πω στην αγαπημόνι μου στην Άλφια ότι δεν ξέρω και σχετικά με τον φόβο που εξέφρασε κατά πόσον είναι αναστρέψιμη η κατάσταση. Ναι, σας λέω ότι δόξα τω Θεώ αναστρέφεται. Μπορεί να αναστραφεί, είναι αναστρέψιμη, αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε για να αναστραφεί να προσπαθήσουμε όλοι μαζί. Ήρθα σε επαφή λοιπόν με τους, ε, τις διάφορες ε, ε, ομοσπονδίες, με εκπροσώπους των διαφόρων θεσμικών οργάνων, τον κύριο Φερνάντο Λόπεθ Μύρας από την περιφέρεια, αλλά και με πολλούς. Για να σας καθησυχάσω, να σας πω ότι πρώτον κατανοώ την ανησυχία σας και εδώ η Κομισιόν όπως μας είπε και ο εκπρόσωπός της γνωρίζει την κατάσταση και γνωρίζει γιατί να σας πω ότι και ο ταπεινός υποφαινόμενος ε, έχει ήδη ζητήσει βοήθεια, εξτραφεί προς την Κομισιόν για να ζητήσει ε, βοήθεια όσον αφορά το θέμα αυτό και πρέπει να συγχαρούμε όλοι τους εαυτούς μας ε, γιατί η Κομισιόν δεσμεύτηκε γραπτά ε, να, δώσει, ε, να στηρίξει με συγκεκριμένους πόρους την περιοχή. Απ' την άλλη πλευρά ε, ε, ε, δεν είναι ένας αυτός που πρέπει να προσπαθήσει. Πρέπει να σας πω ότι η παρούσα κυβέρνηση της Μούρθια έχει ήδη λάβει κάποια μέτρα. Έχει τον, έχει τον νόμο προστασίας του, της Μαρμενόρ, το σχέδιο διαχείρισης της περιφέρειας. Άρα η παρούσα κυβέρνηση της Μουρθία κάνει κάποια πράγματα. Είναι σημαντικό όμως να μιλάμε όχι μόνο για αυτή την πλευρά των πραγμάτων, αλλά και για όλες τις άλλες πλευρές. Και ζητώ, λυπάμαι, λυπάμαι πραγματικά, ε, ε, γιατί... το, ε, η, κεντρική κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικολογικής Μετάβασης ε, ε, ε, είδε ότι σε αυτήν την περίπτωση υπήρχε δημοσιονομική παράλυση. Η το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Μούρθια ήθελε να κινηθεί, αλλά η κυβέρνηση της Ισπανίας θα πρέπει να αποφασίσει να δώσει κάποιους πόρους αφιερωμένους ειδικά για την Μούρθια. Ε, ενώ βλέπουμε ότι δεν υπάρχει τέτοια δημοσιονομική ε, πρόβλεψη ε, ούτε για την περιοχή γενικότερα, ούτε και για τη Μαρ Μενόρ ειδικότερα. Εγώ πραγματικά ήρθα σε επαφή με πολλούς εκπροσώπους και αυτό κατάλαβα. Πάντως σήμερα είμαστε εδώ όλοι εδώ, λέω, για να προχωρήσουμε το θέμα και έτσι ώστε αυτή η υπέροχη λιμνοθάλασσα να επιβιώσει. Αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι πρέπει όλοι να κάνουμε κάτι, όλοι να συμβάλλουμε. Ε, η κυβέρνηση της Μούρθια θα δώσει 56 εκατομμύρια για το ε, πρόγραμμα ε, για την Μούρθια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης, αλλά θα πρέπει να συμμετάσχουμε όλοι για να λύσουμε το θέμα γιατί αυτή η διαδικασία δεν πρέπει να έχει ούτε καμία ιδεολογία, ούτε και οποιοδήποτε πολιτικό χρώμα, μονάχα το γαλανό χρώμα που θέλουμε να έχει η Λιμνοθάλασσα. Ολοκληρώνω κυρία Πρόεδρε λέγοντας το εξής. Σήμερα βρισκόμαστε όλοι εδώ έτσι ώστε να δεσμευτούμε και εγώ σαν Ισπανός υπερήφανος που είμαι για την Ισπανία, υπερήφανος για αυτή τη δικιά μου Μαρ Το έστω και αν δεν είμαι Μουρθιάνος αλλά ε, είμαι από άλλη περιοχή της ε, ε, Ισπανίας, λέω ότι είμαι πεπισμένος ότι όλες οι απειλές και όλοι, όλες οι αμφιβολίες οπωσδήποτε θα λυθούν γιατί θεσμικά ε, έχουμε τις δυνατότητες και οι πολίτες θα βοηθήσουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τους αναφέροντες για τον αγώνα τους και για το γεγονό ότι έφτασαν με τον αγώνα τους μέχρι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχετε αγωνιστεί πάνω από 10 χρόνια ορισμένοι από εσάς και με διάφορες μορφές γιατί το πρόβλημα αυτό δεν είναι καινούριο. Το πρόβλημα της Μαρ Μενόρ δεν είναι κάτι που εμφανίστηκε πρόσφατα, ούτε καν τους τα τελευταία τρία-τέσσερα χρόνια. Είναι πολύ βαθύτερο. Έχει αναφερθεί ότι σε αυτή τη λιμνοθάλασσα έχουμε τη μεγαλύτερη οικολογική καταστροφή σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή. Είναι άνευ προηγουμένου. Και είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει ξεκινήσει και βλέπουμε όλο και νέα επεισόδια. Δηλαδή ξεκινήσαμε από τον ευτροφισμό, ε, φτάσαμε ε, σε ξηρασία, με ανοξία, με διάφορα ε, είδη ψαριών που πέθαναν και έβγαιναν στις ακτές. Και αυτό ξέρουμε πού θα οδηγήσει. Τελικά θα οδηγήσει στην πλήρη εξαφάνιση των ειδών που ζουν σε αυτό το οικοσύστημα, σε μια οικοκτονία όπως λέμε. Υπάρχει οδηγία habitat για τους οικοτόπους και επίσης κάποια άλλα στοιχεία που μας τα δίνει η οδηγία για την προστασία των αγριών πτηνών. Υπάρχει δηλαδή ευρωπαϊκή νομοθεσία. Γι' αυτό ζητούμε να παραμείνει ανοιχτή αναφορά έτσι ώστε να συνεχίσει να παρακολουθεί το θέμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο, αλλά και να, να αναλάβει πρωτοβουλίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κυρίως. Τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει πολύ γοργή τα μεταβολή της χρήσης της γης σε αυτή την περιοχή. Το ανέφερε και η συνάδελφος. Ε, έχουμε εντατική γεωργία, χωρίς έλεγχο, χωρίς σε πολλές περιπτώσεις να ε, γίνεται σεβαστή και η οδηγία για, για τα νητρικά. Είναι η Μούρθια μία από τις ελάχιστες αυτόνομες κοινότητες της Ισπανίας που δεν έχουν σχετικό στρατηγικό σχέδιο για την προστασία του περιβάλλοντος Εμεί γιατί έρχομαι ε, και εγώ, από τη Μούρκια, Μούρθια, είμαστε μία από τι λίγε κοινότητε. μάλλον η μόνη κοινότητα αυτόνομη στην Ισπανία που δεν έχει χώρο ταξικό σχεδιασμό επίση. Εν πάση περιπτώσει, βλέπετε ότι πρόκειται για ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα και οδηγεί και σε οικονομικά προβλήματα και σε κοινωνικά προβλήματα. Γιατί μιλούμε για εκατομμύρια ανθρώπους που επηρεάζονται από το γεγονό ότι δεν μπορούν πλέον να ασκήσουν τι οικονομικέ δραστηριότητε που ασκούσαν όπω είχαν. Όλοι όσοι ζούμε στη Μούρθια με κάποιον τρόπο έχουμε επηρεαστεί ε, περιβαλλοντικά, ψυχολογικά, προσωπικά. Έχουμε κάποιον γνωστό που έχει πληγεί. Ε, ζητώ λοιπόν δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, να ζητήσουμε η Επιτροπή μας να αποστείλει στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, στην ΕΝΒΗ, το αίτημα να οργανωθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια αποστολή διερευνητική. Να επιδιώξαμε και παλαιότερα θυμάστε να οργανώσουμε ως Επιτροπή ε, Αναφορών μια, επιστρο, μια ε, ε, επίσκεψη στη Μαρμενόρ. Δεν έτυχε αυτό υποστήριξη από όλε τι πολιτικέ ομάδε. Εν πάση περιπτώσει ζητούμε αυτή τη στιγμή να γίνει από την ΕΝΒΗ μια αποστολή να υπάρξουν συναντήσει με όλε τι οργανώσει τη κοινωνία των πολιτών, τι περιβαλλοντικέ που αγωνίζονται για, την, για τη Μαρμενόρ και να οδηγηθούμε στη σύνταξη μιας έκθεσης που να περιγράφει την κατάσταση με αποστημονικά δεδομένα και με συστάσεις. Το δεύτερο αίτημα, το οποίο το απευθύνω και προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί ακούσαμε διάφορα από διαφορε προτάσεις, διαφορε ιδέες, εν πάση περιπτώσει, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει πραγματικά ε, μια ε, εμπλοκή τη άμεση, να σταματήσουμε, να, περάσουμε από τα λόγια στι πράξεις, να επισκεφθούν εκπρόσωποι τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής στην περιοχή, να δουν τι συμβαίνει ακριβώ, ε, να, να, δουν πώ είναι πια το νερό, τι χρώμα έχει το νερό στη Μαρμενόρ. λαμβάνουμε πάντοτε αυτές τις δικαιολογίες από την περιφερειακή κυβέρνηση της ε, Μούρθια, ε, όμως πρέπει να υπάρξουν ε, συνέπειες, πρέπει να υπάρξει λογοδοσία. Και ζητούμε λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει τις διαδικασίες τις σχετικές, διαδικασία επί ό,τι χρειάζεται για να αποδοθούν ευθύνες. και θα χρειαστεί τους επόμενους μήνες να καταρτιστούν προγράμματα και να βρεθούν κονδύλια ε, επιπλέον και αυτό το ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα χρειαστεί επιπλέον χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Έχω λοιπόν αυτές, αυτά τα δύο βασικά αιτήματα ε, προς την Επιτροπή ΕΝΒΙ που σας το περιέγραψα, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και φυσικά προς την Επιτροπή μας ζητώ να κρατήσουμε ανοιχτή αυτή την αναφορά. Ευχαριστώ. Thank you. Mr. Weiss, uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν θα επαναλάβω τους επένους για την περιοχή, τι οικολογικός θησαυρό είναι και τι κληρονομιά και για την Ισπανία και την Ευρώπη. Θα σχολιάσω την κατάσταση που αντιμετωπίζουμε. Το πρόβλημα το ξέρουμε εδώ και 30 χρόνια. Προφανώς έχουμε ένα παράδειγμα ε, τοπικών αρχών που είτε δεν θέλουν είτε δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν και να επιβάλλουν ισπανική και νοσιακή νομοθεσία. Εδώ υπάρχει συνειδητή καταστρατήγηση των νόμων που παραβλέπουν οι τοπικές κοινότητες. Οι αγρότες ε, λένε ότι τους επέτρεψαν ή... Ε, τοπικές κοινότητες. Ε, μιλάνε για τα πηγάδια αλλά και τα νητρόδια Αυτά είναι από τη Γεωργία. Και εγώ ε, μπορώ να σας πω ότι μπορεί να είναι κανείς υπεύθυνος αγρότης και με λιπάσματα χωρίς να γεμίζει το έδαφος με νητρόδι και χρειάζονται μεγάλες ποσότητες νητροδών για να πάθει αυτή τη ζημιά η περιοχή. Κανείς δεν μπορεί να μου εξηγήσει πώς γίνεται μετά από τόσα χρόνια και τόσες δεκαετίες να, υπάρχει, να υπάρχουν παράνομα λύματα στο μαρμενόρ χωρίς οι αρχές να παίρνουν χαμπάρι τι γίνεται. Αυτό το παραγνωρίζουν συνειδητά. Η ΠΠΗ είναι συντηρητική στην περιοχή, τώρα έχουμε στην κυβέρνηση τους σοσιαλδημοκράτες και χαίρομαι που ε, και από τους σοσιαλδημοκράτες υπάρχει έκκληση να υπάρξει ενημέρωση και κυρώσεις. Γιατί η διαδικασία έπιβα παραβάση και μάλιστα θετικώς εκπλήσωμε πόσα μέτρα πήρε ήδη η Κομισιόν. Το 2015 παραβάσει ε, ε, ε, παραβάση, κανένα αποτέλεσμα. Το 2017 τίποτα. Γίνονται διάφορα αναφορές, κανένα αποτέλεσμα όμως. Άρα πώς μπορούμε εμείς να εξασφαλίσουμε στους Ισπανούς ότι θα προστατέψουμε το περιβάλλον τους ε, με βάση το Natura 2000. Πρέπει να ανταποκριθούμε αλλιώ. Μην εκπλησώμεθα που δεν πιστεύουν πια στην Ένωση οι πολίτες. Ε, καθήκον μας είναι να φροντίσουμε να αλλάξει η κατάσταση επιτόπου τάχιστα και άρδιν Γι' αυτό έχει δίκιο η Ισπανίδα συνάδελφος, αν νομίζω, να προβλέψουμε συγκεκριμένες ποινές, περικοπές κονδυλίων. Αν στη χώρα μου δεν εφαρμόζονται οι κανόνες και αυτή η διασπορά νητροδών σημαίνει ότι δεν τηρούν οι αγρότες τους κανόνες, τους περικόβεται τις αγροτικές τους επιδοτήσεις, γιατί αυτή τη γεωργία την επιδοτούμε, τη χρηματοδοτούμε. Και ε, συνάδελφος ε, που ε, μίλησε και που εκπροσωπεί την περιοχή πρότεινε μια γεωργική στρατηγική που θα συνεχίζεται χωρίς καμία αλλαγή. Όχι πολύ φιλόδοξη σε ό,τι αφορά την, οργανή, την οικολογική μετάβαση, όχι μείωση των νητροδών. Ε, όχι πολύ οργανική γεωργία. Ε, νητρόδι μπορούν να χρησιμοποιούνται αλλά, ή λιπάσματα, αλλά με τρόπο λογικό. Να πιέσουμε, να περικόψουμε μέχρι να εφαρμόσουν τους κανόνες όπως τους εφαρμόζουν όλοι οι άλλοι αγρότες. Και έτσι νομίζω θα αλλάξουν τα πράγματα, έτσι το βλέπω εγώ, γιατί όταν δουν οι αγρότες ότι δεν παίρνουν επιδοτήσεις πια επειδή δεν φέρονται καλά και δεν τηρούν την νομοθεσία για το έδαφος και το είδωρ, τότε θα δούμε δραματική και άμαση αλλαγή των γεωργικών τους πρακτικών και θα έχουμε θετικό αντίκτυπο στη Μαρ Μενόρ. Ήταν ε, καλή πρόταση από τη συνάδελφα από την Ισπανία ή τη Σοσιαλδημοκρατία. Α πάμε, αν δεν υπάρχει, πάμε αποστολή. Αν δεν υπάρχει πλειοψηφία σε αυτή την επιτροπή, α το θέσουμε στην επιτροπή ένβη. Α πάμε επιτόπου να δούμε, να ελέγξουμε και α ε, τελειώνουμε. Και εγώ παραπονιόμουν για το παρελθόν, αλλά αυτό δεν θα βοηθήσει ούτε το Μαρμενόρ ούτε τους πολίτες εκεί. Επιτέλους, ας αντιληφθούμε ότι τα τελευταία 30 χρόνια δεν γινόντουσαν σωστά τα πράγματα. Να πάμε και να συμβάλλουμε σε μια πραγματική θετική αλλαγή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την συναισθηματικά φορτισμένη αυτή ε, παρέμβαση. Ο κύριος Πενικούβερ. Κύρια Πρόεδρε, Ευχαριστώ πολύ για τις ωραίες παρεμβάσεις. Ευχαριστούμε ε, γιατί πολλά σωστά ελέγχθησαν, γι' αυτό θα είμαι σύντομος. Ευχαριστώ και την Κομισιόν που μας εξήγησε ποια μέτρα θα πρέπει να ε, ληφθούν σε μια περιοχή όπου έγιναν τεράστια λάθη στο παρελθόν και μάλιστα πρέπει να πω και να δώσω δίκιο στη συνάδελφο, δεν αποδίδονται ευθύνες ε, σε σχέση με την τήρηση της νομοθεσίας. Όμως αυτό δεν είναι θέμα μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και οι κοινοτικέ αρχές και η ισπανική κυβέρνηση καλείται να κάνει πολλά βήματα και από κοινού να φροντίσει για λύση του προβλήματος. Εμείς πάντως θέλουμε να διορθώσουμε το οικοσύστημα εκεί. Αυτή είναι η βούλησή μας και η προσπάθειά μας και γι' αυτό πρέπει να προσπαθήσουμε. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει και απλούστευση, αλλά ε, να συνεχίσουμε, να, δώσουμε συνέχεια στην αναφορά την τελευταία του 19. Οι άλλες μπορούν να κλείσουν. Με βάση την τελευταία αναφορά θα ασκήσουμε ε, πίεση στην Κομισιόν ώστε να δώσει περαιτέρω διευκρινήσεις και σε σχέση με το να το δώσουμε στην Ένβη, δεν ξέρω, ίσως θα πρέπει να γίνει μια διερευνητική αποστολή. Μου φαίνεται ότι υπάρχουν και άλλες αναφορές που χρειάζονται βέβαια κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να αναγνωρίσω ότι υπάρχουν άνθρωποι που με καλή πίστη και χωρίς πολιτικές διεκδικήσεις ήρθαν εδώ ε, για να ζητήσουν την ε, επαναφορά της Μενόρ στην αρχική της κατάσταση. Κυρίες και κύριοι, πρέπει να σας πω ότι γνωρίζω από πρώτο χέρι ε, το, την Μενόρ και γνωρίζω τον θησαυρό που η Μενόρ αντιπροσωπεύει. Η πρώτη φορά που τα παιδιά μου είδαν ε, το χρώμα της θάλασσας ήταν ακριβώς στη Μάρ ε, Μενόρ. Εδώ και δύο-τρία χρόνια ε, βλέπω με μεγάλη θλίψη τα όσα συμβαίνουν. Υποφέραμε η οικογένεια, οι φίλοι, οι, οι γείτονες, οι κάτοικοι, όλοι υποφέρουν στη Μαρμενόρ, αλλά υποφέρουν και μέλη της περιφερειακής κυβέρνησης. Εγώ δεν θέλω να υποφέρει κανείς, ε, ούτε και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την πολιτική ε, και τα τελευταία χρόνια Κανείς δεν ήταν ευχαριστημένος. Ωστόσο, εγώ λέω ότι η υπεράσπιση ε, της Μαρ Μενόρ δεν βρίσκεται στα χέρια συγκεκριμένων ανθρώπων και αυτό για ιδεολογικούς λόγους. Οι τοπικές αρχές της Μουρθία βεβαίως ε, ασχολήθηκαν με τα προβλήματα της Μαρ Μενόρ και εξακολουθούν και το κάνουν. Με ικανοποίηση ακούω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που το αναγνωρίζει. Η ε, η περιοχή της ε, Μουρθία μέσω της κυβέρνησής, τους, κυβέρνησής της ε, αναφέρεται στην βιωσιμότητα, στην διερεύνηση, στην ε, ευαισθητοποίηση και σε ένα σωρό άλλα μέτρα. Δεν έχουμε αρκετά χρόνο στη διάθεσή μας για να σας πω ποια είναι τα στοιχεία ελέγχου τα οποία και κυρώσεων που έχει εφαρμόσει η τοπική κυβέρνηση έτσι ώστε να γίνει ε, σεβαστή η ε, οδηγία επίσης ε, όπως ανέφερε και η Κομισιόν, θα μπορούσα να σας μιλήσω για το σχέδιο διαχείρισης του 2019. Πάρα πολλοί είναι αυτοί που συμμετείχαν εις την θέσπιση και τη συγκρότηση αυτού του προγράμματος. Ήδη από, τα από πέρσι υπάρχει συγκεκριμένο μοντέλο Ε, που διαβουλεύεται ε, όσον αφορά τα μέτρα αυτά. Επίσης, ε, πέρσι δόθηκαν πάνω από 8 εκατομμύρια ευρώ και για την Μαρμενόρ 56 εκατομμύρια για, προβλέπονται για διασωτικά και άλλα έργα τα επόμενα χρόνια. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που από ό,τι φαίνεται γράφουν στα παλιά τους υποδήματα αυτά τα στοιχεία. Δεν είναι δυνατόν να πολιτικοποιείται ένα ε, πρόβλημα σαν αυτό της αναβίωσης ε, της ε, Μαρμενόρα. Άκουσα κάποιες δηλώσεις από σοσιαλιστές βουλευτές. Θα ήθελα να θα ήθελα να πω ότι καθόλου δεν στήριξε ο Σάντσες, γύρισε την πλάτη μάλιστα στην περιοχή της Μούρθια όταν ζητούσε βοήθεια. Ε, και όσο και άσχημα να πάει η ε, περιοχή της ε, Μούρθια, ποτέ δεν θα σταματήσει να ασχολείται με την Μαρμενόρ. Για το 1,5 εκατομμύριο των κατοίκων δεν είναι δυνατόν να δεχτούν, να στρέφεται εναντίον του ΕΛΚΑ αυτή η περίπτωση της Μαρ ε, Μενόρ. Ο, η πρόεδρος ε, της ε, περιφέρειας μπήκε σε ένα ελικόπτερο και ε, κοίταξε, είδε πως έχει η κατάσταση. είδε πως έχει η κατάσταση, γύρισε στη Μονκλώα και, και μίλησε με τον Πρωθυπουργό και έδωσαν μηδέν πόρους. Ε, παρα, εξακολουθούν να δίνουν χρήματα στην Καταλωνία, ίσως ε, για να εξαγοράσουν ε, κάποια υποστήριξη στην περιοχή αυτή. Ε, κοιτάξτε, υπάρχουν ε, άνθρωποι οι οποίοι κουνάνε πάντα το δάχτυλο και λένε στους άλλους εμείς είμαστε καλοί, εσείς δεν είσαστε και τόσο. Η χρηματοδότηση από πλευράς ε, της κυβέρνησης δεν ήταν μηδενική, αλλά η περιφέρεια της Μούρθια προσέτρεξε στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έτσι ώστε να ζητήσει δάνειο Ωστόσο, ο Σάντσες απαγόρευσε ε, την ε, ε, έναρξη έργων όσον αφορά την Μούρθια. και το έκαναν αυτό σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών γιατί και παραθέτω η Μούρθια πρέπει να αυξήσει τους φόρους πρώτα πριν στραφεί σε δάνεια. Είναι προφανές ε, ότι ο Πρωθυπουργό ε, της ε, Ισπανίας δεν ενδιαφέρεται ούτε για τη Μούρθια ούτε για την Μαρμενόρα. Ενδιαφέρεται μονάχα για την μικροπολιτική αντιπαράθεση. Εμείς όμως θέλουμε να αφήσουμε πίσω μας την λαϊκίστικη υποκρισία. Ε, θέλουμε να δουλέψουμε όλοι χέρι με χέρι με την κοινωνία των πολιτών, με τους ε, επιστήμονες ε, και δεν πρέπει να αποτελέσει, δεν πρέπει να η κατάσταση της Μούρθια και της Μαρμενόρ και θα πρέπει οπωσδήποτε να μιλήσετε με τον Πρωθυπουργό Σάντσες έτσι ώστε να βάλει και αυτό στο χέρι του για να λυθεί αυτή η πολύ σοβαρή κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Κυρία Αγγελάρμα ε, Γαρθία έχει ζητήσει το λόγο. Αν δεν, έχετε, δεν είχατε πάρει το λόγο. Έχετε πάρει, είχατε πάρει και πριν το λόγο. Μάλλον ο κύριος Ορτασούν. Δεν θέλω να συνεχίσουμε την ε, συζήτηση επί μακρόν, αλλά πιστεύω ότι και η αναφέροντες και η Επιτροπή σε αυτά που μας είπαν κατέδειξαν ότι πιθανώς να έχουν υπάρξει παραβιάσεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας όσον αφορά την προστασία του οικοσυστήματος. Και σε αυτό πιστεύω ότι θα έπρεπε να εστιάσουμε ως Επιτροπή, γιατί το ζήτημα είναι τι μπορούμε να κάνουμε ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας για να βελτιώσουμε την κατάσταση στο Μαρμενόρ. Δεν μου αρέσει αυτή η μικροπολιτική τώρα σύγκρουση που γίνεται μεταξύ ισπανικών πολιτικών κομμάτων. Ε, ας σταθούμε στο σοβαρό πρόβλημα, πρόβλημα που είναι αυτό που μα εξέθεσαν οι αναφέροντε. και να, το ζήτημα είναι να κάνουμε μια συζήτηση που θα οδηγήσει σε λύσεις. Επεβελήθησαν κάποιε προτάσει. Ακούστηκε, για παράδειγμα, να κάνουμε μια αποστολή διερευνητική, να ετοιμάσουμε μια έκθεση. Αυτά μάλιστα, αυτά να τα συζητήσουμε. Αλλά ένα ουσιαστικό σύντημα τώρα που έχει σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος και τη σεβασμό του ευρωπαϊκού δικαίου, παρακαλώ ας μην το ε, εκφυλίσουμε σε μια συζήτηση για τα εσωτερικά πολιτικά προβλήματα της Ισπανίας. Κύριε Αρέγο, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αναφέροντες. Είναι ε, Ιδιαίτερα λυπηρή αυτή η εικόνα που μας ε, φέρνουν οι αναφέροντες με την οικολογική ε, κατακρίμνηση μιας ε, τόσο όμορφης περιοχής. Επίσης θα ήθελα να εκφράσω τη λύπη μου για κάποια από αυτά που άκουσα. Συμφωνώ με τον συνάδελφο Ουρτάσουν ότι εδώ δεν πρέπει να μεταφέρουμε εσωτερικές πολιτικές διαφορές εδώ ε, αντιθέτως ε, συνάδελφοι ε, μίλησαν σωστά συνάδελφοι που πήραν το λόγο προηγουμένως και νομίζω ότι καλό θα είναι αυτή η Επιτροπή να πάει μια αποστολή στη Μαρ για να δει επί τόπου τι συμβαίνει γιατί πραγματικά όταν βρίσκεσαι εκεί στην Μαρ και βλέπεις πως κατάντησε πραγματικά ε, ε, ε, όχι μόνο περιβαλλοντικά αλλά και κοινωνικά και οικονομικά λυπάσαι ειλικρινά αυτά που βλέπουμε, τα στοιχεία που μας ε, φέρνουν ε, ε, όλες οι οργανώσεις αλλά και η επιστημονική κοινότητα, όλα αυτά πρέπει να μας οδηγήσουν στην απόφαση να πάει η Επιτροπή Επιτόπου έτσι ώστε επιτόπου in situ να δει πώς έχουν τα πράγματα. Και βεβαίως όλα αυτά σχετίζονται και με πολιτικές αποφάσεις που ελήφθησαν και από μια συγκεκριμένη κυβέρνηση η οποία πήρε συγκεκριμένες αποφάσεις ε, σύμφωνα με τις οποίες ε, ε, η γεωργία, ναι, ναι, φυσικά νόμιμα, αλλά παρόλα αυτά εξελίχθηκε με τρόπο ώστε να οδηγήσει σε αυτό το πρόβλημα. Ε, και αυτού του είδους οι παράνομες στην ουσία εκμεταλλεύσεις οδήγησαν ε, σε αυτήν την κατάσταση. Όλα θα πρέπει να τα λέμε και χαίρομαι πραγματικά που υπάρχουν άνθρωποι, πολίτες ε, που προβληματίζονται γι' αυτό και γι' αυτό ζητούμε τη στήριξη όλων για να οργανωθεί αυτή η αποστολή. Εμείς λέμε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να μείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά έτσι ώστε να έχουμε έναν μηχανισμό πίεσης για να ληφθούν οι σωστές αποφάσεις και οπωσδήποτε δεν πρέπει ε, να κοροϊδευόμαστε. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο οικονομικό και δεν πρέπει ε, απλώς να βλέπουμε η μία ε, υπηρεσία να στέλνει τον μπαλάκι, να ρίχνει τον μπαλάκι στην άλλη. Χρειάζεται μία πολλαπλή δράση. Όπως είπε και ο συνάδελφος, να γίνει μία αποστολή πρώτον. Δεύτερον, να ασχοληθεί και η Επιτροπή Περιβάλλοντος, η Επιτροπή Έμβη με το θέμα, γιατί όντως είναι συνυπεύθυνη. Επίσης, ε, να ζητήσουμε από τις τοπικές περιφερειακές αρχές να μας εξηγήσουν ποια είναι τα μέτρα τα οποία θα λάβουν έτσι ώστε 15.000 εκτάρια τουλάχιστον παράνομης εκμετάλλευσης στην πεδιάδα της Καρταχένα ε, να ε, σταματήσουν να καλλιεργούνται. Επίσης το γεγονός ότι υπάρχει δυνατότητα αναστροφής εντός των επόμενων χρόνων και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Αγγιλέρα. Ναι, να ξεκαθαρίσω κάτι στο, στο οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Βάης σχετικά με το αγροτικό γεωργικό μοντέλο. Εγώ δεν είπα ότι χωρίς καμία επιφύλαξη ε, ε, συμφωνώ με το μοντέλο γεωργικής ανάπτυξης, λέω ότι τα τελευταία 20 χρόνια δεν ήταν παράνομες οι γεωργικές δραστηριότητες, έγιναν με σύνομο τρόπο. Ε, και ότι επετράπησαν διάφορες διαδικασίες που οδήγησαν σε αυτήν την ε, κατάσταση. Εγώ δεν θέλω να υπεραμεινθώ αυτού του μοντέλου ε, γεωργίας, αλλά από την άλλη μεριά δεν θα πρέπει να θεωρήσουμε ένοχο τον γεωργό. Και να πω το εξής. Εγώ δεν κατάλαβα αυτά που είπε ο συνάδελφος ο Θόιδο όταν ε, λέει ότι ε, δεν θέλω να πολιτικοποιήσω την κατάσταση. Ίσως χρειάζεται μετάφραση αυτών που είπα. Λοιπόν, να μην, ναι, θα δώσω τον λόγο στον κύριο Θόηδο. Ε, για να απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Να ξεκαθαρίσω δύο πράγματα. Πρώτον, έγιναν αναφορές ε, και το ε, ΕΛΚ δεν αντέδρασε, δεν αντιτάχθηκε σε μια ενδεχόμενη αποστολή επιτόπου. Το θέμα ήταν θέμα προτεραιότητας, δηλαδή να υποστηριχθεί Είχαμε πει ότι ε, εμείς κατά προτεραιότητα θέλαμε να, να μελετηθεί το θέμα των 300 και πλέον δολοφονιών της ΕΤΑ που δεν είχαν ξεκαθαριστεί. Εδώ αναφέρονται στο, στο έγγραφο που σας δείχνω όλα τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν από την κυβέρνηση της ε, Μούρθια ε, και οπωσδήποτε θα πρέπει ορισμένοι να προσέχουν και αυτά που λένε και τον τόνο με τον οποίο τα λένε, το ύφος τους. Σας ευχαριστούμε λοιπόν. Θεωρώ ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση εδώ. Και για να ολοκληρώσουμε φυσικά τη συζήτηση θα δώσω στον κύριο Σαλασάρο Ορτούνιο σε δύο λεπτά το λόγο και κύριο Καστεγιάννος άλλα δύο λεπτά, τους αναφέροντες δηλαδή. Αναφέρον. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι το ζήτημα εδώ είναι το εξή. Έχουμε 10.000 εκτάρια τα οποία έχουν ε, καλλιεργηθεί παρανόμως. Γι' αυτό είναι πρόβλημα για όλη την Ευρώπη. Αυτό που ζητούμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι να μας βοηθήσει να εφαρμοστεί το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Όλα αυτά που σας αναφέραμε είναι πράγματα που δεν έχουν συμβεί από τη μια στιγμή στην άλλη και ε, συζητούμε τώρα για νέα νομοθετικά μέτρα ή νέες, νέα, ε, νέους διαλόγους. Ε, η κατάσταση στη Μάρα Μενόρ είναι επίγουσα όμως. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Χωσέ Λουίς ήταν σπάνιο να έχουμε αναφέροντα ο οποίο να, να μην εξαντλήσει το χρόνο του. Κύριε Άλβαρε, έχετε λίγο περισσότερο χρόνο. Εγώ θα ήθελα να υποστηρίξω αυτέ τι προτάσει που ακούστηκαν, δηλαδή να, παραμείνει ανοιχτή, να παραμείνουν ανοιχτέ όλε οι αναφορέ σχετικέ. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό αυτό. Το που συμβαίνει στην ε, Μούρθια δείχνει ότι η κοινοτοποίηση της κοινωνίας των πολιτών μπορεί να οδηγήσει σε προστασία του περιβάλλοντος. Είχαμε κινητοποιήσεις μαζικές στην Καρταγέννη. Και επίσης θα πρέπει να αναλάβει όλες τις πρωτοβουλίες που μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό πιστεύω ότι είναι απολύτω απαραίτητο. Αν θέλουμε να βρεθεί μια κάποια λύση για αυτά τα προβλήματα της Μαρμενόρ, χρειάζεται να ε, είναι η πίεση στις τοπικές αρχές. Το πρόβλημα είναι πολύ απλό Δυστυχώ. Έχουμε ένα μοντέλο ε, οικονομικό και παραγωγής αγροτικής το οποίο καταστρέφει το περιβάλλον. Δηλαδή, τα δύο μοντέλα που έχουμε για την προστασία, το μοντέλο για την προστασία του περιβάλλοντο και το οικονομικό μα μοντέλο δεν είναι συμβατά μεταξύ του. Άρα, εάν δεν αλλάξει το μοντέλο το οικονομικό τη Καρθαγέννη, δεν πρόκειται ποτέ να προστατεύσουμε αυτό το οικοσύστημα στη Μαρ Μενόρ. Εάν θέλουμε να παραμείνει εν ζωή το οικοσύστημα στη Μαρμενόρ, είναι απολύτω απαραίτητο να αλλάξει ο τρόπο με τον οποίο γίνεται η γεωργία σε αυτή την περιοχή. Ε, η συντριπτική πλειονότητα των ε, ε, λιμάτων και των, των βαρέων μετάλλων προέρχονται από αυτέ τι δραστηριότητε. Σα ευχαριστούμε. Μετά λοιπόν από την συζήτηση και την ακρόαση και των αναφερόντων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η πρόταση της Προεδρίας είναι να παραμείνει η αναφορά ανοιχτή. Επίσης, να ζητήσουμε πληροφορίες από το ε, Υπουργείο Οικολογικής Μετάβασης Περιβάλλοντος της Ισπανίας για στοιχεία, για μέτρα που έχουν ληφθεί για την προστασία ε, της Μαρ Μενόρ, για ε, την γεωργική παραγωγή στην περιοχή και στοιχεία για τον προϋπολογισμό σχετικά. Θα ζητήσουμε σχετικά στοιχεία από την Περιφερειακή Κυβέρνηση της Μούρθια να μας αναφέρει τι μέτρα και τι πόρους έχει δώσει και κατά τη διάρκεια του 2018-19. Επίσης θα ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή περισσότερες πληροφορίες Ήδη έχουμε αρκετά στοιχεία ως ε, Επιτροπή Αναφορών, αλλά θέλουμε ακόμα περισσότερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πιο συγκεκριμένα θέλουμε να μας δώσετε επενδυτικά σχέδια που να έχουν εγκριθεί ή να έχουν υποβληθεί από τις περιφερειακές αρχές της Μαρμενόρ για την προστασία την περιβαλλοντική της περιοχής. Επίσης, η Επιτροπή μας θα ζητήσει από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, την ΕΝΒΗ, ε, την διοργάνωση μιας διερευνητικής αποστολής στην περιοχή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους πολίτες της Ισπανίας που ήρθατε εδώ στο... Ε, στον οίκο της δημοκρατίας, αν θέλετε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εδώ που μπορείτε να εκφράσετε τη φωνή σας. Σας ευχαριστούμε που αναδείξατε και αναδεικνύετε διαρκώς το θέμα αυτό και ε, θα προσπαθήσουμε να σας υποστηρίξουμε στις προσπάθειές σας και στις προσπάθειές μας να βελτιώσουμε την κατάσταση του περιβάλλοντος στη Μαρ Θα προχωρήσουμε τώρα στο σημείο 11 της ημερήσιας διάταξης. Ο κύριος H.E. από τη Γερμανία, εκπροσωπώντας την ομάδα πίεσης Trilander Region Gegen Tiange, στο συγγνώμη για την προφορά, και το ζήτημα συζήτησης είναι ο πυρηνικός σταθμός του Τιχάνγκε. Καλώς ορίσατε ένα πραγματάκι μόνο να σας ζητήσω ε, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Θα ήθελα να ζητήσω, να από τους ε, από να αποχωρήσουν ησύχω. Περνάμε στην επόμενη αναφορά. Πέντε λεπτά θα σας δώσω και στο τέλος θα έχετε και δύο λεπτά ακόμα για να κλείσετε. Παρακαλώ, έχετε το λόγο και καλώς ήρθατε. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Αναφορών, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής. Έχει περάσει ένας χρόνος από τότε που ήρθα για το τυχόν εξ ονόματος του Δήμου του Άχεν τότε είχαμε ζητήσει περισσότερες πληροφορίες και θέλαμε και να απευθυνθεί επιστολή στη βελγική κυβέρνηση. Από τότε δυστυχώς δεν έγινε τίποτε από την Κομισιόν και έτσι πρέπει να επαναλάβω τις κατεπίγουσες εκκλήσεις μας. Ε, ο Δήμος του ε, Άχεν και οι τρεις περιοχές ε, περιφέρεια τριών χωρών κατά του Τιχάνς ε, από το Λουξεμβούργο και την Γαλλία. Ε, θα ήθελα να αναφερθώ στον πυρηνικό σταθμό Τιχάνς 2, για τον οποίο υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες. Τον Ιούλιο του 19, ο πυρηνικός αντιδραστήρας ε, άρχισε πάλι να χρησιμοποιείται μετά από χρόνια όπου δεν λειτουργούσε. Τον Οκτώβριο, λόγω τεχνικών προβλημάτων, έπρεπε πάλι να σταματήσει. Σοβαρές ε, αμφιβολίες ε, υπάρχουν από το 2012 σχετικά με τη λειτουργία του και την ασφάλειά του. Το 2012 για πρώτη φορά σταμάτησε. Υπάρχουν ρογμές. Το, τα αίτια δεν έχουν ακόμα, των ρογμών αυτών δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί. Οι βελγικές αρχές το 2013 παρόλα αυτά αποφάσισαν την επαναλειτουργία. Το 2014 μας είπε ο επιχειρηματίας ότι ο, ο ε, είπε ότι οι ρογμές ήταν μεγαλύτερες από ό,τι είχαμε αρχικά θεωρήσει. Σταμάτησε πάλι. Έγινε έκθεση ε, μετά από έρευνα ε, οι αμφιβολίες δεν διασκεδάστηκαν και το Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 2015 άρχισε πάλι να λειτουργεί ο πυρηνικός αντιδραστήρας Τιάνς 2. Ε, πολλοί ανεξάρτητοι επιστήμονες, ειδικοί, ειδικές επιτροπές αμφισβητούν την ε, ασφάλεια του σταθμού. Επίσης υπάρχουν και άλλες ε, περιπτώσεις ε, δηλώσεων δυσλειτουργιών στην, που αφορούν τις τρεις χώρες Ολλανδία, Λουξεμβούργο και Γερμανία. Εν τω μεταξύ και στο χώρο ασφαλείας του αντιδραστήρα διαπιστώθηκαν ε, προβλήματα και ανομαλίες. Ε, έχει ε, υποστεί ζημία το μπετόν που, χρησιμοποιείται, που χρησιμοποιήθηκε για το καταφύγιο. Ε, λόγω δημιουργίας καυτού ατμού που διαχρονικά πέδρασε αρνητικά στο μπετόν για την διασφάλιση του σταθμού θα πρέπει το καταφύγιο αυτό να μπορεί να είναι απόλυτα ε, λειτουργικό. δεν ε, γνωρίζομαι αν μπορεί να ανταποκριθεί σε εξωτερικές, ε, εξωτερικά προβλήματα για παράδειγμα, αν μπορεί να ανθέξει σε περίπτωση ε, κατάρριψης αεροσκάφους. Ε, είναι σημαντικό να εξεταστούν όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν το σταθμό Τιχάνς 2, ε, τα οποία δεν έχουν παρόλες τις εκκλήσεις υποβληθεί. Η Επιτροπή Αναφορών καλείται κατεπηγόντως προς υποστήριξη, ούτως ώστε να μπορέσουμε να διερευνήσουμε τα δεδομένα του σταθμού. Οι βελγικές αρχές θα πρέπει να μας υποβάλουν και να μας τεκμηριώσουν ε, τα στοιχεία περί της ασφάλειας. Επίσης, ε, θα πρέπει να ε, διατυπωθεί αίτημα απέναντι προς το βασίλειο του Βελιγίου. Τα στοιχεία που δεν έχουν ακόμα υποβληθεί πρέπει να δοθούν. Το βασίλειο του Βελγίου θα πρέπει να εγγυηθεί για τα περίπου 8 εκατομμύρια κατοίκων που θα επηρεαστούν αρνητικά σε περίπτωση προβλήματος του Τιχάνς 2. Επίσης καλείται η Επιτροπή και τη νέα Επιτροπή ε, να, την, ε, ε, να ζητήσει από τη νέα Επιτροπή να ε, εξετάσει την αρχή προφύλαξης και πρόληψης σε σχέση με τον πυρηνικό σταθμό τη 2. Ευχαριστώ. Και τώρα η Κομισιόν. Ε, δεν είστε αναφέρον, ναι. Ο Βάλτερ Σούμαχαρ. Α, που είναι αναφέρον. Εγώ ε, προέρχομαι από πρωτοβουλία των πολιτών κατά των πυρηνικών. Συμφωνώ με τα όσα είπε ο προηγούμενος ομιλητής, εμείς θέλουμε κι άλλα στοιχεία, θέλω να παρακολουθήσουμε, να δούμε τι κάνουν οι αρχές ε, ασφάλειας, υπεύθυνες για την ασφάλεια στο Βέλγιο, τι έγγραφα έχουν, τι έρευνες έχουν κάνει. Αν είχαμε όλα αυτά τα έγγραφα, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε μια πολύ καλή δουλειά και ανάμεσα στις οργανώσεις βάσης, αλλά και σε επιστημονικό και πολιτικό επίπεδο. Ε, συνεχίζουμε λοιπόν να επιμένουμε. Φροντίστε κι εσείς οι βελγικές αρχές να μας δώσουν τα απαραίτητα έγγραφα. Σας ευχαριστώ. Και τώρα η Κομισιόν, η Ανέτα Σιέσκα. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Κυρία Πρόεδρε, Ευχαριστώ, ευχαριστώ και τους αναφέροντες για τις παρουσιάσεις και τις ανησυχίες που εκδήλωσαν. Καταρχήν η Κομισιόν και πάλι τονίζει ότι καταλαβαίνει και παρακολουθεί τις ανησυχίες που εκφράζονται από τους πολίτες σχετικά με την ασφάλεια του πυρηνικού σταθμού Χάνς 2. Η πυρηνική ασφάλεια και η προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος είναι απόλυτες προτεραιότητες της Κομισιόν. Η Κομισιόν θα ήθελε να επαναλάβει ότι οι αποφάσεις σχετικά με την ασφάλεια αυτών των σταθμών είναι θέμα κρατών μελών. Και η ε, υπεύθυνοι ε, για την, ε, να φροντίσουν για την ασφάλεια είναι η υπεύθυνη λειτουργία του σταθμού που υποβάλλουν τις εκθέσεις τους. Για το νομικό, ρυθμιστικό πλαίσιο έχει ε, μετατεθεί στο Εθνικό Δίκαιο ή Οδηγία για την πυρηνική ασφάλεια. Τώρα συνεχίζουμε για να δούμε αν όλες οι συνιστώσεις, όλα τα στοιχεία της οδηγίας έχουν μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία με τρόπο σωστό και επίσης επαληθεύομαι και βελτιώνομαι ε, με προτάσεις στα θέματα ασφάλειας. Εκτός αυτού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ομάδα των ρυθμιστικών αρχών οργάνωσε την πρώτη επανεξέταση ε, στα πλαίσια της οδηγίας για την πυρηνική ασφάλεια. Το Βέλγιο συμμετείχε στην άσκηση αυτή. Ε, η έκθεση ε, από τους ομοτήμους έγινε, αξιολόγηση έγινε και ήδη τα αποτελέσματα έχουν δημοσιευτεί το, στο τέλος του 2018. Τον Νοέμβριο του 2018 έγινε συνάντηση στις Βρυξέλλες και το έργο συνεχίζεται. Τα κράτη-μέλη θα έπρεπε να προετοιμάσουν ε, εθνικά προγράμματα δράσης σχετικά με τις ε, που αφορούν τα ειδικά ευρήματα για την κάθε χώρα τον Σεπτέμβριο του 2019 υπευλήθησαν τα εθνικά σχέδια. Το Βαέλγιο επίσης υπέβαλε το εθνικό σχέδιο. Υπάρχουν αυτά στην ιστοσελίδα και ε, όπως και οι δράσεις που απαιτούνται από τα κράτη-μέλη. Εκτός αυτού τον Νοέμβριο του 2019 ε, η ΕΝΣΡΕΓ e δέχτηκε ένα συνολικό πρόγραμμα δράσης εκτός από τα εθνικά. Υπάρχει και αυτό στην ιστοσελίδα της ΕΝΣΡΕΓ. E Ο στόχος του προγράμματος δράσης είναι να παρακολουθούμε τις ε, οδηγίες ε, με βάση τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί και να αρχίσει η νέα διαδικασία αξιολόγησης από τους ομοτήμους, γιατί αυτό συνεχίζεται. Στο τέλος του Μαΐου του 2021 οι διεθνείς ρυθμιστικές οι αρχές θα πρέπει να κάνουν μια ενημέρωση του προγράμματος δράσης. Και τα επόμενα βήματα είναι τα ενημερωμένα εθνικά προγράμματα που θα χρησιμοποιηθούν για να καταρτιστεί μια συνολική έκθεση της ENSREG. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Ο κύριος Αβι... Αχιμών. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκρούτε Μάιερ εξήγησε γιατί είμαστε ακόμα εδώ και πιέζουμε. Εγώ είμαι στο, από τη βελγική πλευρά, 20 χιλιόμετρα μακριά από εκείνον. Είμαι δηλαδή πολίτης αυτού του κράτους που εξακολουθεί να διατηρεί και να λειτουργεί το πυρηνικό σταθμό. Όμως προσυπογράφω και με τα δύο χέρια όσα είπε. Έχω ασχοληθεί ε, πολύ με το θέμα αυτό και έχω μιλήσει και με ειδικού που εξακολουθούν να αμφιβάλλουν ε, αν λόγω των αμφιβολιών που υπάρχουν και εξακολουθούν να υπάρχουν για τον πυρηνικό σταθμό αν μπορεί αυτός να λειτουργεί. Ίσως ε, θα έπρεπε να περάσει από δοκιμή ένα κομμάτι του σταθμού. Αλλά είναι δύσκολο να δούμε αν αυτός ο πυρηνικός αντιδραστήρας μπορεί να ανθέξει ε, εξωτερικές πιέσεις. Δύσκολο αυτό να γίνει αν δεν λειτουργεί. Όλες αυτές οι δοκιμές είναι δηλαδή που έχουν γίνει, μάλλον θεωρητικές είναι και μόνο. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ατυχήματα, γι' αυτό νομίζω ότι όλες οι πληροφορίες ε, που έχει η Βελγική Ομοσπονδία για την Πυρηνική Ασφάλεια και τον Πυρηνικό Έλεγχο όλες τις πληροφορίες που έχει να τις διαθέσει στους αναφέροντες που να δώσει και την αξιολόγηση από τους ομοτήμους και όλα τα σχετικά, ούτω ώστε να εξεταστούν από ειδικού. Εγώ έλαβα γνώση σχετικά με την η υλοποίηση της σχετικής οδηγίας από το 87 που ε, προβλέπει ότι πρέπει να υπάρχουν αμοιβαία αξιολογήσεις από ομοτήμους μεταξύ των κρατών μελών που θα λαμβάνουν υπόψη και τη διαχείριση της ε, απαρχαίωσης των ε, πυρηνικών αντιδραστήρων είναι ένα καλό πρώτο βήμα ούτως ώστε να έχουμε μια ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας για τα πυρηνικά. Πήγα στο Λουξεμβούργο και απευθύνθηκα ε, σε ειδικού ε, της αρμόδιας αρχής, ε, μηχανικούς, που εξετάζουν κάθε μέρα τα θέματα πυρηνικής ασφάλειας και εκεί εκφράστηκε μια επιθυμία και είναι και ερώτημα προς την εκπρόσωπο της Κομισιόν και παράκληση η Ευρώπη σχετικά με την πυρηνική ενέργεια συνεργάζεται, αλλά όχι σε ό,τι αφορά το θέμα της ασφάλειας των πυρηνικών αντιδραστήρων. Αυτό, όπως ελέγχθη πολύ σωστά, εξακολουθεί να είναι αποκλειστικά εθνική αρμοδιότητα. Παρόλο που υπάρχουν οι αξιολογήσεις απομοτήμους, υπάρχει εθνική αρμοδιότητα. Αυτή η βελγική αρχή, λοιπόν, είναι η μόνη που μπορεί να αποφασίσει αν παρά τις επιφυλάξεις που υπάρχουν σχετικά σε ολόκληρη την Ευρώπη μπορεί να αποφασίζει αν θα συνεχίσει να λειτουργεί όχι το πυρηνικό σταθμός. Μόνο αυτή. Έτσι έχει το πράγμα. Καλός ή κακός. Δεν θα το συζητήσουμε. Η πυρηνική ενέργεια όμως και οι βιομηχανικές διαδικασίες που στηρίζονται από εκεί ε, είναι διασυνοριακά θέματα, γιατί αν έχει πρόβλημα ένας αντιδραστήρας, θα έχουν πρόβλημα και άλλες χώρες. Δεν μπορεί να... Δεν υπάρχει όμως μια Ευρωπα... ένας ευρωπαϊκός οργανισμός που αν υπάρχουν επιφυλάξεις θα αναλάβει να εξετάσει το θέμα και θα δει σε ευρωπαϊκό επίπεδο αν πρέπει ένας αντιδραστήρας να κλείσει ή όχι. Οι οργανισμοί ε, δεν καλύπτουν όλα τα προβλήματα και το έχω δει. Οι άνθρωποι στην περιοχή είναι πάρα πολύ φοβισμένοι ε, σχετικά με τις ειδήσει που ακούνε από το Τιχάντζε. Είναι κρίμα που δεν υπάρχει ένας τέτοιος οργανισμός. Εγώ απευθύνω έκκληση στην Κομισιόν να τα σκεφτεί όλα αυτά και να δει αν ή τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να συμφωνήσουν υπέρ μια, της ίδρυσης ενός ευρωπαϊκού οργανισμού γιατί είναι πυρηνική ασφάλεια στα πλαίσια της συνθήκης της Ευρατόμ. Να μην ε, κρεμόμαστε μόνο από την απόφαση του βελγικού φορέα. Και θα πρέπει παρακαλώ να κρατηθεί η αναφορά ανοιχτή μέχρι να πάρουμε όλα τα στοιχεία και να μπορούμε και εμείς με τους δικούς μας ειδικού να ε, διαμορφώσουμε γνώμη. Ευχαριστώ. Κύριος Φρόιντ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ο συνάδελφος ε, μίλησε πολύ ξεκάθαρα. Ο πυρηνικός αντιδραστήρας είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα, γιατί αν συμβεί κάτι, σε αυτή την περίπτωση τέσσερις χώρες τουλάχιστον πλήττονται και παρόλα αυτά μια χώρα δικαιούται να αποφασίζει αν θα μείνει στο δίκτυο ο πυρηνικός αντιδραστήρας. Γι' αυτό πολύ σωστά απευθυνθήκαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τώρα θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, ούτω ώστε τα θέματα που άπτονται της πυρηνικής ασφάλειας, των κινδύνων ασφαλείας των ε, αντιδραστήρων να ε, απαντηθούν ικανοποιητικά. Το Βέλγιο ε, δεν επιτρέπεται να αγνοεί τις αμφισβητήσεις, τις αμφιβολίες μας και να συνεχίζει απρόσκοπτα. Η Κομισιόν θα πρέπει στα πλαίσια του Ευρατών να ε, προχωρήσει στις αρμοδιότητες που έχει για τον έλεγχο. Τα τελευταία χρόνια είδαμε με πολύ παράδοξο τρόπο ότι στο Τιχάνς μια ανοίγουν, μια κλείνουν τον αντιδραστήρα, αρχίζουν τα προβλήματα, τα ψευτοδιορθώνουν και αρχίζει, αρχίζουμε πάλι από την αρχή. Το θέμα είναι πάρα πολύ ε, λεπτό έχει να κάνει με την πυρηνική ενέργεια. Η αδιαφάνεια επιβάλλεται και ο πληθυσμός στη Γερμανία, στην Ολλανδία, στο Βέλγιο και στο Λουξεμβούργο σε αυτή την περίπτωση έχει δικαίωμα να γνωρίζει σε ποιους κινδύνους ακριβώς είναι εκτεθειμένοι. Η συνθήκη Ευρατών που την αναφέραμε ρυθμίζει τα θέματα πυρηνικής ασφάλειας στην Ευρώπη αλλά είναι ένα μαύρο κουτί αυτό. Όχι ότι δεν ε, έχουμε εποπτεία με οργανισμό, αλλά είναι ένας από τους λίγο τομείς όπου δεν έχουμε και κοινοβουλευτικό έλεγχο. Από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας όλοι οι άλλοι τομείς ήταν υπό τον έλεγχο των, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά στην Ευρωατόμ εδώ και 60 χρόνια δεν έχει υπάρξει καμιά αλλαγή ούτε και έλεγχος. Μετά το Brexit ούτως ή άλλως θα πρέπει να ξανανοίξουμε τη συνθήκη αυτή και είναι τώρα καλή ευκαιρία και για μας και, και, και εμείς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σκεφτούμε την αναθεώρηση της ε, Euratom και να προβλέψουμε και τέτοιο οργανισμό και να δούμε και τον, τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε και το ρόλο της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Γερμανίας γιατί ε, τροφοδοτεί το ΤΙΑΝΣ ε, με στοιχεία καύσης και νομίζω ότι ήρθε η Γερμανία να βγει απ' έξω και να μην δίνει το υλικό καύσης για τον ε, αντιδραστήρα. Σε τακτά διαστήματα γίνονται διαδηλώσεις από τους πολίτες ενάντια στον αντιδραστήρα. Μην τους εγκαταλείψουμε. Οι βελγικές αρχές χθες το βράδυ, λίγες ώρες πριν έρθουμε εδώ, μετά από ένα χρόνο, κούνησαν το δαχτυλάκι τους και απάντησαν στην επιστολή από αυτή την Επιτροπή. Αλλά δεν υπάρχει απάντηση στην επιστολή που ε, έστειλαν. Είπαν ότι εμείς είμαστε πεπισμένοι ότι είναι ασφαλεί οι αντιδραστήρε και να μας εμπιστεύεστε σε αυτά που σας λέμε. Έτσι όμως δεν οικοδομείται εμπιστοσύνη. Οι αναφέροντες και εμείς θέλουμε αυτά τα έγγραφα που αφορούν τις ασφάλειες να δοθούν, να εξεταστούν από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και εσείς ε, και νομίζω ότι ως Επιτροπή Αναφορών πρέπει να απευθύνουμε επιστολή στην Κομισιόν και να καταγράψουμε ποια έγγραφα έχει πάρει ήδη η Κομισιόν και αν αυτά επιτρέπουν έναν έλεγχο ασφαλείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επίσης η Επιτροπή Αναφορών θα πρέπει να ε, απαντήσει στο γράμμα το χτεσινό από το Βέλγιο και να ζητήσει όλες τις αναλύσεις ε, για την ασφάλεια που θα δοθούν στην, πρέπει να δοθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να γίνει ανεξάρτητος έλεγχος. Γιατί δεν μπορεί αυτοί που λειτουργούν το σταθμό να αυτό πιστοποιούνται και να λένε ότι όλα είναι εντάξει. Ελπίζω ότι με αυτά θα γίνει πιο γρήγορη η εξέλιξη και να μην χρειαστεί να περιμένουμε πάλι ένα χρόνο μέχρι να μας απαντήσουν. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν η Κομισιόν θέλει να απαντήσει στην ερώτηση του Ευρωβουλευτή Αριμών. Η Κομισιόν θέλει να ευχαριστήσει τον αναφέροντα για τα σχόλια. Τα έχω σημειώσει βεβαίως Προς το παρόν περιορίζομαι μόνο σε αυτή τη δήλωση. Ευχαριστώ. Ωραία. Τώρα, δύο λεπτά έχετε για το κλείσιμο. Ο κύριος Ρουτεμάιερ, Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Υπενθυμίζω αυτό που αποφάσισε η Επιτροπή πριν από ένα χρόνο. Είχε, πει, είχε αποφασίσει ότι καλεί την Κομισιόν για περισσότερες ε, πληροφορίες και η ε, Επιτροπή θα συνεχίσει την αναφορά στο βαθμό που δεν έχει λάβει τις απαραίτητες πληροφορίες. Ακούσαμε πρόσφατα ότι αυτές οι πληροφορίες μέχρι τη σημερινή ημέρα δεν έχουν δοθεί και η δήλωση της Κομισιόν δεν συνέβαλε στη διαφάνεια και στο ξεκαθάρισμα, οπότε παρακαλώ να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά ε, και όπως ε, ζήτησε και ο Ευρωβουλευτής Αριμών, να εκφραστεί η, η παράκληση, να δοθούν όλα τα έγγραφα για να γίνει συζήτηση επί τη βάση αυτών των εγγράφων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σούμαχερ. Δεν θέλετε? Δεν θέλετε. Ε, Ευχαριστούμε πολύ όλους τους αναφέροντες που για την παρουσία τους ακούσαμε την αναφορά, ακούσαμε τις απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις τοποθετήσεις των συναδέλφων. Η πρόταση της Προεδρίας είναι να παραμείνει αναφορά ανοιχτή, να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλη την τεκμηρίωση και όλα τα στοιχεία που μπορεί να μας δώσει Επίσης, να ζητήσουμε πληροφορίες από τη βελγική κυβέρνηση όλα τα στοιχεία που έχουν σχέση με την ασφάλεια αυτού του πυρηνικού αντιδραστήρα. Η Επιτροπή Αναφορών επίσης θα ζητήσει ε, και η ίδια από την βελγική κυβέρνηση τα στοιχεία αυτά. Δηλαδή ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τα ζητήσει από το Βέλγιο και εμείς θα τα ζητήσουμε απευθείας από το Βέλγιο επίσης. Και η αναφορά παραμένει ανοιχτή. Ευχαριστώ. Θα συνεχίσουμε τώρα με το σημείο 12 τη ημερη διάταξη. Πρόκειται για την αναφορά που θα παρουσιάσει ο κύριος Λουσιάν Σαουλένου από τη Ρουμανία, 690 του 2018, εκ μέρου τη Ένωσης για την Αναγέννηση της Κράιοβα σε σχέση με την πρόταση να ε, δοθεί παράταση στη λειτουργία του πυρηνικού αντιδραστήρα Κοσλοντούι στη Βουλγαρία. Βλέπω ότι παρίσταται ο αναφέρον. Έχετε λοιπόν 5 λεπτά για να μας παρουσιάσετε την αναφορά σας. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, εγώ είμαι ο εκπρόσωπος της 784, είναι αναφέρον 784. Θέλετε να συνεχίσω, ωραία. Μπορούμε να εξετάσουμε λοιπόν την 784 πρώτη. Κοιτάξτε, στο σημείο 12. συγγνώμη, εγώ έκανα λάθος, λέει πρόεδρο. Λοιπόν, στη 12 πράγματι έχουμε δύο αναφορέ. Την 690 του 2018 του κυρίου Σάου Λένου από τη Ρωμανία και επίση την 784 του 2019 ε, που θα την παρουσιάσετε εσεί ε, από τη Βουλγαρία. Εκπροσωπείτε επίση και μία ε, μη κυβερνητική οργάνωση Βούλγαρων και Ρουμάνων πολιτών για τα προβλήματα από τα ραδιενεργά απόβλητα. Δεδομένου ότι ο πρώτο αναφέρον δεν παρευρίσκεται, θα δώσω σε εσά το λόγο για πέντε λεπτά για να μα παρουσιάσετε τη δική σα αναφορά. Ελάτε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ενημερώσω ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία ε, στην αναφορά μας που έχουν αλλάξει. Που έχουν ε, ε, νέες εξελίξεις. Για, μάλλον πιο σωστά. Το ζήτημα της αναφοράς στο, με το οποίο προσπαθούμε να, στο οποίο προσπαθούμε να αναφερθούμε είναι η δημιουργία ενός αποθετηρίου για τα απόβλητα τα πυρηνικά που δημιουργεί ο πυρηνικός αντιδραστήρας Κοσλοντούι, ε, το οποίο θα προτίθενται να εγκαταστήσουν στη Βουλγαρία. Έγιναν συναντήσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και των Βουλγαρικών Αρχών και της ε, Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας της Βουλγαρίας, που είναι αρμόδια και για την ε, συγγνώμη, την ε, ρυθμιστική αρχή για την πυρηνική ενέργεια στην Βουλγαρία, που είναι αρμόδια και για την ε, ρύθμιση των αποθητηρίων πυρηνικών αποβλήτων. Έχει αναγνωριστεί ότι υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά τη στατικότητα αυτής της περιοχής που βρίσκεται κοντά στο Δούναβι. Πρόκειται για μια περιοχή όπου το έδαφος δεν είναι, είναι σαθρό, δεν είναι σταθερό το οποίο σημαίνει ότι μπορεί να, αν δημιουργηθεί εκεί αποθετήριο, θα έχουμε παραβίαση της οδηγίας για την διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων. Και... Πιο συγκεκριμένα, συγκεκριμένων ισοτόπων που έχουν ε, αυξημένη ημιζωή. Μιλάμε για ισότοπα, ορισμένα από αυτά έχουν η ζωή που ξεπερνάει τα εκατομμύρια, κάποιες χιλιάδες χρόνια. Το ζήτημα λοιπόν που τίθεται είναι, εάν έχει γίνει σωστά η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αναφέρονται μόνο ε, ισότοπα τα οποία έχουν μικρή ημιζωή. Θεωρούμε λοιπόν ότι υπάρχει κίνδυνος παραβίασης της οδηγίας του 2011 που ρυθμίζει τη διαχείριση των, περιβα... των ραδιενεργών αποβλήτων. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχει έλλειψη διαφάνειας στη Βουλγαρία όσον αφορά την αδειοδότηση και τη λειτουργία ε, εγκαταστάσεων πυρηνικής ενέργειας. Είναι κάποια συγκεκριμένα πολιτικά κόμματα εκείνα που προωθούν τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας στη χώρα μου. Εδώ όμως δεν μιλάμε για τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας. Μιλάμε για κάτι πιο συγκεκριμένο. Μιλούμε για απόβλητα τα οποία είναι επικίνδυνα και τα οποία, και, γίνονται ακόμα πιο επικίνδυνα αν σκεφτούμε ότι θα αναποτεθούν σε μια περιοχή η οποία ε, έχει προβλήματα ε, στο έδαφος, ε, σταθερότητα στο, του έδαφους. Οι μελέτες είχαν βασιστεί μόνο σε κάποιες προκαταρκτικές αξιολογήσεις Επομένω, εμένα η αίσθηση που μου δίνεται είναι ότι οι τοπικέ αρχέ απλώ προσπαθούν να απορροφήσουν ευρωπαϊκού πόρου και να απορροφήσουν και του πόρου από το ειδικό ταμείο για, την, για το Κουσλοντούι. Αλλά α μην ξεχνούμε ότι αυτά τα χρήματα είναι χρήματα των Ευρωπαίων φορολογωμένων. Ζητούμε λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ελέγξει ε, πιο αυστηρά την κατάσταση να ελέγξει τι συμβαίνει ακριβώς. Βλέπετε αυτή τη στιγμή στην οθόνη έναν πίνακα τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν θα επηρεάσουν πολλές γενιές. Σας το είπα, η ζωή αυτών των αποβλήτων είναι τεράστια κάποιον από τα ισότυπα που συμπεριλαμβάνονται σε αυτά τα απόβλητα. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι ένα πρόβλημα που θα επηρεάσει πολλούς ανθρώπους σε βάθος χρόνου. Ελπίζουμε λοιπόν ότι θα γίνει μια ανεξάρτητη αξιολόγηση, αναθεώρηση αυτών των μελετών Έχουμε ήδη επιστημονικά στοιχεία που δείχνουν ότι η περιοχή αυτή είναι ασταθής. Η πρόεδρο διακόπτη πρέπει να ολοκληρώσετε σιγά σιγά. Α, ε, ολοκληρώσατε. Εντάξει, ευχαριστώ. Τέλεια. Θα δώσω το λόγο στην Κομισιόν η κυρία Αντουανέτα Ζωβακαλάπης. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον αναφέροντα που ήρθε. Είναι πράγματι πολύ ανησυχητικά όλα αυτά που φοβάται. Όμως το Εθνικό Δικαστήριο ασχολήθηκε εκτενώς με αυτό το θέμα γιατί η απόφαση εμφισβητήθηκε στο δικαστήριο και το δικαστήριο διατήρησε την απόφαση. Η Κομισιόν δεν έχει λόγο να αμφιβάλλει τα συμπεράσματα του δικαστηρίου που λέει ότι οι ανησυχίες των αναφερόντων δεν τεκμηριώνονται. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τη συνθήκη για την, ε, τη συνθήκη Ευρατόμ και με βάση τα γενικά δεδομένα που έδωσε τα κράτη-μέλη σχετικά με τα ραδιενεργά κατάλοιπα, η Κομισιόν αποφασίζει αν ένα τέτοιο ε, ένα σταθμός μπορεί να οδηγήσει σε ρήπανση δάφους ε, νερού σε ένα άλλο κράτος μέλος. Το Δεκέμβριο η Κομισιόν εξέδωσε απόφαση και είπε ότι το ε, πρόγραμμα δεν είναι... Ε, δεν θα οδηγήσει σε ραδιενεργό μόλυνση ενός άλλου κράτους μέλους, η εθνική δηλαδή εγκατάσταση διάθεσης ραδιενεργών αποβλήτων. Η Κομισιόν ζήτησε τη βοήθεια ειδικών εμπειρογνωμόνων για τη ραδιενέργεια. Όπως προβλέπει η συνθήκη, η ομάδα αποτελείται από ειδικού στο θέμα της ραδιενέργειας και η Κομισιόν δεν έχει λόγο να αμφισβητήσει την εμπειρογνωμοσύνη του σε σχέση με αυτό. Να προχωρήσουμε την επόμενη αναφορά. Τώρα, για την ε, άλλη, ε, την αναφορά του 2019, ότι δεν έγινε καλή οργάνωση για να ε, εξεταστεί η ασφάλεια, η Πέρσι τον Ιούλιο είχε γίνει η πρώτη απάντηση. Η Κομισιόν δεν είδε ελλείψη στη διαδικασία των διαφουλεύσεων σε σχέση με το διασυνοριακό αυτό έργο. Η προσέγγιση των ε, ορισμένων μερών ε, ήταν ε, επιπόλαιοι και ε, η, πρώτα, η, η, άποψη αυτή υπάρχει στην ιστοσελίδα μας και στις ιστοσελίδες της ε, βουλγαρικής και ρουμανικής κυβέρνησης. Επίσης, εξηγήθηκε σε σχέση με την άλλη αναφορά του 18 ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι βουλγαρικές ή ρουμανικές αρχές έχουν παρεκκλίνει από το εφαρμοστέο ενωσιακό ή διεθνές δίκαιο. Επίσης, η Βουλγαρία έχει κάνει όλα τα βήματα για να ενημερώσει τη Ρουμανία τον Μάρτιο του 2014, ε, τρεις μήνες πριν ε, κυρωθεί η συνθήκη για την ασφάλεια. Επαναλαμβάνω ότι δεν υπάρχουν διαδικαστικές παραβιάσεις των σχετικών οδηγιών σε αυτή την περίπτωση. Γι' αυτό η Κομισιόν δεν προτίθεται να δώσει συνέχεια στα θέματα που τίθενται σε, αυτήν την, σε αυτές τις αναφορές. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Σλαβάκοφ. Ευχαριστώ. Ίσως ε, εγώ θα ε, κάνω έτσι πιο συναισθηματικό λόγο. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει γκλάσνοστ, διαφάνεια περιβαλλοντική και άλλη. Γιατί πρέπει να σας πω ότι ο πατέρας μου δεν υπέφερε την πρώτη περιβαλλοντική οργάνωση στην ε, Βουλγαρία και τούτη η κατάσταση είναι πολύ επικίνδυνη. Έχω εδώ τη γνωμοδότηση της Επιτροπής ε, Περιβαλλοντική Διαφάνεια, Environmental Glasnost, ε, που εδώ αναφέρεται ως περιθωριακή οργάνωση. Με προβληματίζει πάντως το γεγονός ότι το να λέει να αναφέρεται κανείς στο περιβάλλον ή σε ακτιβιστές για το περιβάλλον είναι σχεδόν κακή λέξη. Από ό,τι φαίνεται πολλοί πιστεύουν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα όσον αφορά ε, τις, ε, την απόρριψη ε, λιμάτων και ε, τη διαχείρισή τους και φαίνεται ότι τα προβλήματα ε, ε, γιατί λένε ότι οι ακτιβιστές αν πάρουν χρήματα μπορούν να πούνε οτιδήποτε. Δηλαδή αν είχαν πάρει χρήματα για να πούνε τι ωραίο που είναι η εγκατάσταση θα το είχαν πει. Ε, σας το βάει είμαι. Κοιτάξτε, εγώ Πράγματι, με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτή ε, η, οικολογική διαφάνεια και λυπάμαι που μερικοί καταστρατηγούν αυτές τις αρχές και βεβαίως θέλω να κλείσει αυτή η, ε, οδηγή, ε, αυτή η αναφορά. Ο κύριος Δαμπάσκη, ευχαριστώ πρόεδρε. πραγματικά με σοκάρει αυτή η πολύ άσχημη και κακόβουλη ε, ε, επίθεση ε, σε αυτό τον σταθμό πυρηνικής ενέργειας. Προηγουμένως μιλούσαμε για βελγικούς σταθμούς, αλλά όταν μιλάμε για το Κοσλοντούι αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο συζητούμε. Ναι, ε, έχουμε τώρα να αντιμετωπίσουμε περιβαλλοντικά ζητήματα, έχουμε να αντιμετωπίσουμε την νέα πράσινη ε, συμφωνία και πραγματικά εκπλήσωμε που μερικές βουλγαρικές ε, οργανώσεις είναι εναντίον αυτής της, του Κοσλοντούι. Ίσως ε, τους ενδιαφέρει μονάχα ε, να υπερασπίζονται τα δικά τους συμφέροντα. Ε, και φαίνεται ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι θύματα ελλειπούς περίθαλψης, υγειονομικής περίθαλψης. Υπάρχουν επίσης άνθρωποι με ε, προβλήματα νοητικά στις, ε, στο, στις, στη Βουλγαρία. Είναι χώρα που, και διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ε, παίρνουν χρήματα, συμβάσεις κλπ. Από την άλλη μεριά έχουμε τους εμπειρογνώμονες ε, που μελέτησαν αυτήν την ε, αναφορά. Αυτή η έκθεση ε, βρίσκει απέναντί της τους λεγόμενους πράσινους ε, ακτιβιστές. Κοιτάξτε, η ιδέα για τη δημιουργία ενός εθνικού αρχείου ξεκίνησε πριν από καιρό σε συνεργασία ή μάλλον βάση των εθνικών και διεθνών αρχών. και συμπεριλήφθη ε, και η οδηγία του 11 καθώς επίσης και όλα τα νομοθετήματα τα οποία αφορούν ε, την ε, ε, υπεύθυνη διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων καθώς επίσης και όλων των στοιχείων που προβλέπει ο Οργανισμός Πυρηνικής Ενέργειας. Σε εθνικό και διεθνές επίπεδο έγιναν σεβαστά όλα τα πρότυπα. Ε, αυτό το αρχείο, το repository, έχει στόχο върху околната среда и човешкото здраве. Целта на оценката на въздействието върху околната среда, освен... Ε, συγγνώμη, αυτό το αποθετήριο έχει ε, αποτελέσει αντικείμενο πρώτερης ε, μελέτης επιπτώσεων στο περιβάλλον. Ε, και έχει ελεγχθεί το ε, σωστό του περιβαλλοντικό ε, καθεστώς, η αντίστασή του και η αντοχή του απέναντι σε ατυχήματα και καταστροφές. Και άλλωστε υπάρχουν και πολλά έγγραφα τα οποία λαμβάνουν υπόψη την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων που έχει γίνει βάσει των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντως, όλη η διαδικασία της εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων απορρέει από το ευρωπαϊκό δίκαιο. Έχει γίνει σωστά και άλλωστε ε, συνάδουν με αυτά οι αποφάσεις του Εθνικού Δικαστηρίου ε, στην ε, Βουλγαρία. Η διαφάνεια της ε, διαδικασίας επομένως ε, είναι δεδομένη και αναγνωρισμένη. Αναγνωρίζεται επίσης ε, ότι η διαδικασία εκτίμησης επιπτώσεων έχει λάβει χώρα βάσει των σωστών στοιχείων και με τον δέοντα τρόπο. Η δε ε, αποφάσεις και εκτιμήσεις έχουν δεόντως κοινοποιηθεί. Θα πρέπει να μην λησμονούμε ότι έχουν γίνει διαβουλεύσεις. Κοιτάξτε, όχι τόσο γρήγορα, γιατί βλέπετε έχουμε τους διερμηνείς εδώ που ταλαιπωρούνται. Ναι, δεν έχουμε και πολύ χρόνο συνήθως γι' αυτό. Ναι, θα τα λέω πιο αργά. Έλεγα λοιπόν ότι θα ήθελα να σας ζητήσω να λάβετε υπόψη το γεγονός ότι και στη Βουλγαρία αλλά και στην Ρουμανία έχουν γίνει ε, δημόσιες διαβουλεύσεις ε, και δεν υπήρξε καμία αντίθετη γνώμη των αρμοδίων αρχών. Θα ήθελα να πω ότι αυτές οι λεγόμενες αναφορές στην ουσία δυναμητίζουν τις διαδικασίες οι οποίες ε, ε, καθοδηγούνται από σωστές εκτιμήσεις επιπτώσεων και επιτρέπουν επενδύσεις σε αυτές τις εγκαταστάσεις. Ποιες είναι αυτές ε, οι δήθεν ε, περιβαλλοντικές οργανώσεις. Ποιοι είναι οι στόχοι ε, που επιδιώκουν. Θέλουν απλά να σταματήσουν ένα project το οποίο σχετίζεται με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Βουλγαρία όσον αφορά τις πυρηνικές εγκαταστάσεις συμπεριλαμβανομένου και ε, του υπεύθυνου τρόπου διαχείρισης των ραδιενεργών αποβλήτων. Εδώ λοιπόν έχουμε μία αναφορά η οποία ε, δημιουργεί πρόβλημα στην Βουλγαρία αλλά και ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα έπρεπε εδώ υπάρχουν συγκεκριμένες αποφάσεις ε, των δικαστηρίων και δεν είναι δυνατόν να επιτρέπουμε ε, σε οποιονδήποτε να ε, υπονομεύει τις διαδικασίες και τις αποφάσεις. Υπάρχουν όλα τα τεκμήρια και τα αποδεικτικά στοιχεία που δείχνουν ότι θα πρέπει να σταματήσει η μελέτη αυτής της αναφοράς και να κλείσει. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Ευχαριστώ. Θα μιλήσω και εγώ στα βουλγαρικά. Και θα πω ότι ως εκπρόσωπος των σοσιαλδημοκρατών οποιαδήποτε υποψία που αφορά την ασφάλεια των πολιτών ε, πάντοτε λαμβάνεται πάρα πολύ σοβαρά υπόψη. Εμείς πρέπει να συμμορφωνόμαστε με τις ε, νομοθεσίες τις ευρωπαϊκές και τις εθνικές. Η έκκλησή μου είναι να κλείσει η αναφορά. Αλλά ως βουλγαρός ε, υπήκος και σοσιαλιστής είμαι κατά οποιασδήποτε προσπάθειας να γίνει η πολιτική ενέργεια ε, αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης. Ευχαριστώ ευχαριστούμε. Ο κύριος Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Συνάδελφοι, σίγουρα δεν συμφωνώ με τη, γνωμοδότηση, με τη γνώμη των αναφερόντων σχετικά με τον πυρηνικό, το πυρηνικό εργοστάσιο του Κοσλοντούι και την εγκατάσταση διάθεσης ραδιενεργών αποβλήτων. Η Βουλγαρία ενημέρωσε τη ρουμανική κυβέρνηση σχετικά με την παράταση του κύκλου των αντιδραστήρων 5 και 6 και παρουσιάσαμε και απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις που έθεσε η ρουμανική κυβέρνηση με το παραπάνω. Εν ώψη της δράσης της Κομισιόν πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει λόγος να πιστέψουμε ότι υπήρξε παραβίαση κανόνων. Για το είναι κατάσταση διάθεσης δεν είναι μόνο προτεραιότητα για τη Βουλγαρία, είναι και δέσμευση. Η Βουλγαρία ανέλαβε τη δέσμευση αυτή ενώπιον της Κομισιόν σε σχέση με τον παροπλισμό των ε, αντιδραστήρων 1 με 4 ε, και αυτό συνάδει με τις προϋποθέσεις ασφαλείας ε, ε, καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων. Ε, είναι η οδηγία του 2011 και αφορά και αυτό το σημείο. Επίσης, βάση της βουλγαρικής νομοθεσίας των προτύπων ασφαλείας του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, διαχείριση αποβλήτων μέχρι το 2030. Όλα, όλες οι νομικές νομοθετικές προϋποθέσεις είναι στη θέση τους και ε, συμμορφωνόμαστε προς αυτές και σε σχέση με το περιβάλλον, την ε, προστασία από την ακτινοβολία των ανθρώπων και του περιβάλλοντος. Τώρα για την εγκατάσταση διάθεσης έγινε ε, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων καταρχήν σύμφωνα με τον, την Εθνική Νομοθεσία και την ε, Σύμβαση ε, για τα διασυνοριακά. Πολλές συζητήσεις επίσης έγιναν και στη Βουλγαρία και στην Κραϊόβα, στη Ρουμανία. Υπάρχει μια συμφωνία πλαίσιο για διάλογο μεταξύ των δύο χωρών. Το 2016 στη Ρουμανία έγινε μια ακρόαση και τέθησαν 23 ερωτήσεις από τους Ρουμάνους πολίτες. Οι βουλγαρικές αρχές έδωσαν πάντοτε γραπτές ερωτήσεις. Και το 2017 δόθηκαν λεπτομερέστατες πληροφορίες από τη Βουλγαρία σχετικά με την κατασκευή αυτής της εγκατάστασης διάθεσης παράλληλα με, επιτροπέ, με ομάδες εμπειρογνωμόνων η Κομισιόν κατέληξε ότι η εγκατάσταση διάθεσης δεν ε, απειλεί καμία χώρα, ε, κατ' ουδένα τρόπο. Και αυτό επιβεβαιώνεται από την ε, έκθεση ε, εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων πάνω σε αυτή τη βάση η αποφάσισε να μην αναλάβει περαιτέρω δράση κατά της Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Εν ώψη όλων αυτών πιστεύω ότι πρέπει να κλείσουν οι αναφορές διότι επειδή υπάρχουν όλες αυτές τις πληροφορίες, μπορούμε να πούμε ε, ότι ε, μπορεί να παραταθεί και να παραταθεί η ζωή των αντιδραστήρων και στην εγκατάσταση διάθεση ραδιενεργών αποβλήτων πληρώθηκαν όλες οι προϋποθέσεις και η Κομισιόν άλλωστε στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξε. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Μπορώ να μιλήσω στα δανεικά. Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε. Εμένα με εξέπληξε λίγο ή και πολύ ε, ο τρόπος με τον οποίο διεξήχθη αυτή η συζήτηση, αυτά που άκουσα. για τα πυρηνικά απόβλητα υπάρχει τεράστια ανησυχία στους πολίτες της Δανίας, είναι γνωστό αυτό. Και γνωρίζουμε ότι δύσκολο, είναι μια τεράστιο πρόβλημα να βρεθεί πού θα αποτίθενται αυτά τα ραδιενεργά απόβλητα. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για όλε τι χώρε. Και ξαφνικά μα λένε οι Βούλγαροι συνάδελφοι ότι το έχουν λύσει αυτό το πρόβλημα. Ότι εκείνοι ξέρουν ακριβώ πού θα εναποθέτουν τα πυρηνικά του απόβλητα και με ένα μαγικό τρόπο όλα πάνε καλά. Λοιπόν, ε, αντιλαμβάνομαι ότι αυτή τη στιγμή στην Επιτροπή μας, επειδή έχουν μείνει μόνο οι Βούλγαροι συνάδελφοι, ή με μάλλον μειοψηφία, αλλά Πιστεύω ότι το θέμα αυτό πρέπει να μας ε, ε, επασχολήσει σοβαρά, ότι θα πρέπει να παραπέμψουμε την αναφορά στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα ακούγοντας και την τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πάλι είναι ξεπλάγινη, γιατί και πάλι ε, η θεωρία ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και φυσικά μεγάλες χώρες όπως η Γερμανία και άλλες θα επιθυμούσαν να βρεθεί μια λύση για το ζήτημα των πυρηνικών απροβλήτων που παράγουμε στην Ευρώπη. Έχουμε όμως πολίτες Ευρωπαίους οι οποίοι έχουν αξιοποιήσει ένα νομικό εργαλείο που τους δίνουμε, ένα θεσμικό εργαλείο μάλλον που τους δίνουμε για να μας εκφράσουν τις ανησυχίες τους εδώ, την Επιτροπή Αναφορών, θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε τις αναφορές τους με σοβαρότητα, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ζήτημα που έχει σχέση με την ασφάλεια των πολιτών. Γιατί δεν τα πιστεύω αυτά. Είναι καταπληκτικά τα πράγματα στη Βουλγαρία. Ξαφνικά, αν όλοι στείλουμε τα πυρηνικά μα απόβλητα στη Βουλγαρία, δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Βρήκαμε τη λύση. Λοιπόν, ζητώ να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά και να την παραπέψουμε στην Επιτροπή Περιβάλλοντο. Παρακαλώ, όχι διάλογο. Κύριο Ναμπάκοφ. Συγγνώμη, συνάδελφοι. Νομίζω ότι τα ραδιενεργά απόβλητα δεν έρχονται όλα στη Βουλγαρία. Δεν ξέρω ποιος σας είπε ότι όλα τα ραδιενεργά απόβλητα πάνε για διάθεση στη Βουλγαρία. Να τελειώσω. Ήθελα να σας πω ότι Ίσως δεν γνωρίζετε αρκετά για πυρηνικού, πυρηνικά εργοστάσια παραγωγής ενέργειας. Δηλαδή, σας είπε κανείς ότι τα απόβλητα της Δανίας θα πάνε στην Βουλγαρία. Αυτά είναι παράλογα πράγματα, όπως είναι και η αναφορά. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, ίσως να υπήρξε πρόβλημα στην διερμηνία. Αλλά από ό,τι είδα κάποιου άλλου συναδέλφου, τα πρόσωπά του μάλλον καταλάβαιναν, εν πάση περιπτώσει. Κοιτάξτε να δείτε, θα απαντήσω. Εσεί είπατε ότι είναι απολύτω ασφαλέ. Και λέω εγώ, αφού στη Βουλγαρία είναι όλα τα πράγματα έτσι λιμένα και είναι απολύτω ασφαλή, ε, γιατί να με στείλουμε και άλλε χώρε τα απόβλητά μα στη Βουλγαρία. Αλλά το λέω με ηρωνία, προφανώ και δεν πιστεύω ότι υπάρχει ασφάλεια. Αυτή είναι η κατάσταση. Ευχαριστώ. Разбира се, колежки, може да складираме вашите стига да платите. Благодаря ви. Βέβαια. Βέβαια, αν χρειαστεί μπορούμε να φροντίσουμε για τη διάθεση αποβλήτων από τη χώρα σας, αλλά θα πληρώσετε. Ωραία, ευχαριστώ. Για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση, θα δώσω το λόγο στον αναφέροντα για δύο λεπτά. Благодаря. Μόνο να γελάσει κανείς μπορεί με αυτή την πολιτική μάχη. Θέλω να διευκρινίσω ότι είμαι αντιπρόεδρος ενός εθνικού κινήματος που λέγεται τη οικολογική διαφάνεια. Όχι ο πολιτικός οργανισμός. Και η οδηγία αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο στη Βουλγαρία. Και λέει ότι η εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα γίνεται από ανεξάρτητο φορέα και στην περίπτωση αυτής της εγκατάστασης διάθεσης και αναφέρομαι μόνο σε αυτή την εγκατάσταση ανεξάρτητη εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων έγινε από μια εταιρεία που παίρνει όλα τα πυρηνικά έργα. Λέγεται Risk Engineering και χρηματοδοτεί όλους τους πολιτικούς. Για μισό λεπτό, κύριε Αλεξάνδροφ. Ολοκληρώνεται λοιπόν η συζήτηση. Ολοκληρώνεται η συζήτηση. Έχοντας ακούσει την Κομισιόν, τον αναφέροντα τους βουλευτές, ε, μέλος, ε, ε, μέλη διαφόρων πολιτικών ομάδων. Η πρόταση της, οδηγή, της Προέδρου είναι να κλείσει η αναφορά καθότι η Κομισιόν καθό, είπε ότι δεν παραβιάζεται οτιδήποτε και κανένα δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα να κλείσουμε αυτή την αναφορά. Um, the, micro. We didn't Sorry. Sorry. Διαμαρτύρομαι γιατί δεν υπάρχει απαρτία. Προτείνω λοιπόν να το συζητήσουμε στους συντονιστές, γιατί τέτοιες αποφάσεις δεν είναι δυνατόν να λαμβάνονται με τόσο λίγα πλήρη μέλη παρόντα. Δεν είναι δυνατόν εδώ να μιλάμε με μέλη που δεν είναι μέλη και που προέρχονται όλοι από την ίδια χώρα. Δεν νομίζω ότι είναι αξιοπρεπή σε αυτή η διαδικασία. Εν πάση περιπτώσει, αν επιμένετε, τι να σας πω. Ωστόσο, δεν είναι ένας ε, σωστός τρόπος ε, για να αντιμετωπίζει κανείς ε, τους αναφέροντες. Πρόεδρος, με γνωρίζετε, ξέρετε ότι εγώ είμαι πάντα δίκαιη. Άκουσα προσεκτικά. Ακούστε με λίγο, κυρία Όουκεν. Ακούστε με λίγο. Προσπαθώ να ολοκληρώσω, να κλείσω τη συζήτηση. Με γνωρίζετε πολύ καλά. Ξέρετε ότι οι αποφάσεις μου και οι συζητήσεις μου είναι σωστές. Άκουσα ε, τους ε, αναφέροντες ε, και ε, ε, βεβαίως τους δώσαμε το λόγο γιατί πάντα η πόρτα αυτής της Επιτροπής Αναφορών είναι ανοιχτή και αποτελεί και πορεία εισόδου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επρόκειτο για ένα θέμα το οποίο προηγουμένως μελετήσαμε, εξετάσαμε ένα θέμα αντίστοιχο για τον αντιδραστήρα Τιάνς του Βελγίου και εδώ ακούσαμε και μας είπαν ότι δεν υπάρχει κάποια παραβίαση ε, δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ Ακούσαμε στην προκείμενη περίπτωση εκπροσώπους του ECR, ε, το, του ΕΛΚ, των Πρασίνων και των Σοσιαλιστών ε, ε, και οι περισσότεροι ζήτησαν να κλείσει η αναφορά συμφωνώντας ή έχοντας ακούσει τα όσα είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν υπάρχει δηλαδή κάποια παραβίαση ενωσιακού δικαίου. Κοιτάξτε, και έχουμε αρκετά μέλη. Και εγώ άλλωστε είμαι μέλο τη επιτροπή. Ακούσαμε προσεκτικά εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων, ακούσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ε, σύμφωνα με αυτά που είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η πλειοψηφία των εκπροσώπων των πολιτικών ομάδων απεφάνθησαν ότι θέλουν να κλείσει η αναφορά. Δεν νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει λόγος να ε, συνεχίσουμε. Άρα, απλώς συνεχίζουμε με το επόμενο, ε, ολοκληρώνουμε τη συζήτηση, κλείνουμε την αναφορά και προχωράμε. Περνάμε στο σημείο 13. Πρόκειται για την αναφορά 827 του 2018 της κυρίας Όλγας Δασκάλη, ελληνική ηθαγένεια, σχετικά με εικαζόμενε σοβαρέ παραβιάσεις των μαθησία Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη διαδικασία διαδότηση τεσσάρων σταθμών ηλεκτροπαραγωγή σε μια προστατευόμενη φυσική περιοχή του Δήμου Μεσολογγίου που βρίσκεται στην Ελλάδα. Νομίζω ότι η κυρία Όλγα Βασκάλη ε, είναι εδώ. Πολύ ωραία. Καλώς ορίσατε κυρία μου. Έχετε πέντε λεπτά στη διάθεσή σας έτσι ώστε να αναφερθείτε στο θέμα. Παρακαλώ έχετε το λόγο. Σα ευχαριστώ πολύ. Έρχομαι σήμερα από το Μεσολόγγιο Λοκαρνανίας. Είμαι δικηγόρο και πρόεδρο του Συμβουλίου Κοινότητα Μεσολογγίου. Άκουσα πριν με πολύ ενδιαφέρον και προσοχή τα προβλήματα που υπάρχουν και στη Μούρθια τη Ισπανία και τώρα πρόκειται να σα πάω σε μια άλλη λιμνοθάλασσα που βρίσκεται στην Δυτική Ελλάδα. Πρόκειται για τον δεύτερο μεγαλύτερο υγρότοπο ε, της, Ανατολικής Μεσογείου, τη δεύτερη μεγαλύτερη λιμνοθάλασσα της Ευρώπης, από τους σημαντικότερους προορισμούς στην Ευρώπη για bird watching. Μιλάμε για μια έκταση πάνω από 300.000 στρέμματα και θα ήθελα να γνωρίζετε ότι η περιοχή αυτή συγκαταλέγεται στους 11 διεθνούς σημασίας υγροβιότοπους της συνθήκης Ραμσάρ, έχει καταχωρηθεί στη ζώνη ειδική προστασίας για τα πουλιά, έχει χαρακτηριστεί ειδική προστατευόμενη περιοχή με τη σύμβαση Τη της Βαρκελόνης, περιλαμβάνεται στον κατάλογο περιοχών του δικτύου Natura, τμήματα του υγροτόπου έχουν χαρακτηριστεί ως διατηρητέα μνημεία της φύσης και καταφύγια θυραμάτων, ενώ μέσα στο Εθνικό Πάρκο υπάρχει και το βιογενετικό απόθεμα του δάσους του Φράξου. Ποιο είναι το πρόβλημα και γιατί βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Μέσα σε αυτό το Εθνικό Πάρκο που προστατεύεται από όλα τα παραπάνω, χωροθετήθηκαν μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιορευστών εντός του κάμπου του Ευνοχωρίου σε απόσταση αναπνευστικής αναπνοής από τη Λιμνοθάλασσα εντός πλημμυρικής ζώνης της λεκάνης του ποταμού Εβίνου με δίκτυ δυνητικής πλημμύρας υψηλό. Η χωροθέτηση αυτή παραβιάζει κατάφορα το άρθρο 11 της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί παραβλέπει τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής. Συγκεκριμένα, το σχέδιο ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης, το βασικό δηλαδή περιφερειακό εργαλείο σχεδιασμού και ανάπτυξη μια περιοχή, στην περιοχή μας προωθεί τη γεωργία, την κτηνοτροφία, την αλληλεία, καθώς επίσης και την ήπια οικοτουριστική ανάπτυξη ανάπτυξη. Πώς μπορεί όμως να επιτευχθεί αυτό όταν μέσα σε αυτή την περιοχή της της αγροτικής παραγωγής σημασίας χωροθετούνται βιομηχανικές μονάδες παραβλέπονται ξεκάθαρα οι αρχές της πρόληψης και της προφύλαξης του άρθρου 191 της συνθήκης αφού η κεντρική διοίκηση εσφαλμένα επιτρέπει να αδειοδοτηθούν βιομηχανικές μονάδες μέσα στην προστατευόμενη περιοχή χωρίς να υπάρχει μελέτη που να δικαιολογεί τους λόγους εγκατάστασης των μονάδων χωρίς να έχει συνταχθεί ειδική οικολογική αξιολόγηση χωρίς να υπάρχει στην περιοχή μας τοπικό χωριστικό σχέδιο με χρήση γης και παρουσιάζοντας μία μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων με παραπλανητικά στοιχεία. Σας λέω απλά χαρακτηριστικά ότι ένας μέσος άνθρωπος διαβάζοντας τη μελέτη βλέπει ότι αναφέρεται σε άλλη περιοχή η οποία βρίσκεται 140 χιλιόμετρα από εμάς, μιλά για τον κάμπο ως ορεινό όγκο, παρουσιάζει μια μελέτη διασποράς ρήπων μιας εβδομάδας ενώ χρειάζεται τουλάχιστον μελέτη ετήσια, μιλά για θέσεις εργασίας όταν τα συστήματα είναι αυτοματοποιημένα και δουλεύουν μόνο ένα με δύο φύλακες. Έχουμε μια κατάφορη εξαπάτηση απάτηση και εσκεμμένη σύγχυση, διότι ξεκινούν παίρνοντα άδεια για να καύσουν βιομάζα, στη συνέχεια όμω με τρει τροποποιήσει πηγαίνουν στα βιορευστά. Αλλάζουν δηλαδή εντελώ την πρώτη ύλη και την μεθοδολογία. Η, η αεριοποίηση τη βιομάζα δεν παράγει βιοαέριο, αλλά συνθετικό αέριο. Στη μελέτη ταυτίζουν το συνθετικό αέριο με το βιοαέριο, κάτι που είναι εντελώ αντιπιστημονικό. Επίση, κατασκευάζουν διάσπαρτα τέσσερι μονάδε στην ίδια περιοχή για να σπάσουν την ισχύ ε, με σκοπό να αποφύγουν την άδεια λειτουργία από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργεια, την άδεια παραγωγή και το επιχειρηματικό σχέδιο και αλλάζουν καθοριστικά το τοπίο τη λιμνοθάλασσα. Επίση, παραβιάζεται κατάφορα και εξόφθαλμα η σύμβαση του Άρχου. Πρέπει να γνωρίζετε ότι στην περιοχή μα δεν υπήρξε καμία διαβούλευση, καμία γνωμοδότηση, καμία ουσιαστική ενημέρωση. Οι πολίτε το έμαθαν όταν τα εργοστάσια άρχισαν να χτίζονται. Δεν προλάβαμε να ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μα. Έτσι δημιουργήθηκε μια έντονη αντίδραση και κοινωνικά κινήματα από φορεί τη πόλη, ο Δήμο Μεσολογγιού, οι τοπικέ κοινότητε, σωματεία εργαζομένων, το τεχνικό επιμελητήριο, δικηγορικό σύλλογο, πολιτιστικοί σύλλογοι, άτυπε ομάδε στράφηκαν εναντίον αυτή τη βιαιότητα. Το ίδιο συμβαίνει να γνωρίζετε και σε άλλε περιοχέ τη Ελλάδα. Επομένω, πρέπει να ξέρετε ότι αυτή την αναφορά σήμερα την υποστηρίζουν ο Δήμο Μεσολογγίου και όλοι ανεξαιρέτω οι φορεί τη περιοχή. Υπάρχει μια αιμονή τη διοίκηση στην Ελλάδα, παραβιάζοντα τη συνθήκη ε, την οδηγία, με συγχωρείτε, 28 του 2009, η οποία ενώ σαν φιλοσοφία έχει την ενημέρωση και την προτροπή για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μας δημιουργούν με μια τέτοια λάθος χωροθέτηση μια αντιπροπαγάνδα κατά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στην περιοχή μας υπήρξαν πάρα πολλέ παρεμβάσεις συγκεντρώσεις, φτάσαμε μέχρι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, εκεί καταφέραμε να αλλάξει νομοθεσία, όμως αυτή η νομοθεσία δεν είχε αναδρομική ισχύ για εμάς. Πρέπει να γνωρίζετε ότι τα τελευταία 20 χρόνια έχουν δαπανηθεί στην περιοχή περιοχή μας πάνω ε, από ε, πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ που προέρχονται από προγράμματα εδαφικής ε, συνεργασίας. Σας αναφέρω χαρακτηριστικά το πρόγραμμα BIG, Συνεργασία Ελλάδας-Ιταλίας, που έχουν να κάνουν με θέματα διαχείρισης και... just one more minute. Ναι. Έχουν λοιπόν χαλαστεί πολλά χρήματα από ευρωπαϊκά κονδύλια και έχουμε τώρα μια εγκληματική αμέλεια και μια αστοχία τη διοίκηση να ακυρώσει όλε αυτέ τι προσπάθειε. Ο τοπικό πληθυσμό ζει μέσα από την, ιχθυοπαραγωγή ενώ οι νέοι άνθρωποι θέλουν να ζήσουν μέσα από την αγροτική παραγωγή και την ήπια οικοτουριστική ανάπτυξη. Εγώ έρχομαι σήμερα εδώ εκπροσωπώντα μια γενιά που έχει παραλάβει ένα σημαντικό υγρότοπο διεθνού σημασία. Θέλουμε να τον προστατέψουμε. Αν δεν ανακληθούν αυτέ οι άδειε, μπαίνει ακόμα ένα λιθαράκι στην υποβάθμιση του περιβάλλοντός μας. Υπάρχει ομόφωνη απόφαση από όλους τις φορείς της περιοχής. Πλέον γνωρίζετε κι εσείς, σας έχουμε φέρει και καινούργια στοιχεία ε, που ε, δείχνουν ότι η αναφορά αυτή θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να προστατεύσουμε και να αναπτύξουμε τον τόπο μας με σχεδιασμό, με λογική και σεβασμό για το οικοσύστημα. Μας έκανε εντύπωση η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την οποία τη θεωρούμε θεματοφύλακα της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, μιας νομοθεσίας που στη συγκεκριμένη περίπτωση παραβιάζεται κατάφορα. Ευχαριστώ πολύ και ζητάμε από εσά να λάβετε άμεσα μέτρα για να αρθούν οι άδειε και ε, με, το να μείνει ανοιχτή αναφορά να δοθεί πίεση στην ελληνική διοίκηση να διακόψει τι εργασίε και εκ βάθρων να επανεξεταστεί η αδειοδότηση. Ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη για τον παραπάνω χρόνο. Κομισιόν. Πολ Σπάιτ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και την αναφέρουσα. Αυτή η περίπτωση είναι μεμονωμένη περίπτωση κακής εφαρμογής. Έχουμε ένα χώρο που δεν έχει να κάνει με πρόβλημα συμμόρφωσης, δεν έχει να κάνει με διαρθρωτικό πρόβλημα στα κράτη-μέλη. Η Κομισιόν παρακολουθεί τις πληροφορίες που παίρνουμε από τις μεμονωμένες καταγγελίες, έχουμε τους καταγγέλλοντες και έχουμε και τις αναφορές. Αλλά όπως είπαμε σαφώς στην ανακοίνωση της Κομισιόν και τις εσωτερικές κατευθυντήριες γραμμές που τη συνοδεύουν και που δεσμεύουν κάθε υπηρεσία της Κομισιόν και του περιβάλλοντος, δεν χρησιμοποιούμε ε, προηγούμενες ε, ανακοινώσεις ή πιλωτικά σχέδια για να κάνουμε την εξέταση. Εδώ, για να κρίνει, θα έπρεπε, θα έπρεπε το Εθνικό Δικαστήριο, το Εθνικό Κράτος Μέλος και μου φαίνεται έχουν γίνει κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση και υπάρχουν δύο είδη. Υπάρχει μη λειτουργικό ε, νοσιακό δίκαιο Οπότε αυτό είναι για το Συμβούλιο της Ευρώπης τον Εθνικό Δικαστή ή ο Εθνικός Δικαστής ε, όπως προβλέπεται η συνθήκη είναι ο αρμόδιος για να κρίνει τα θέματα αυτά. Θα μπορούσε να είναι το Συμβούλιο Επικρατείας. Ε, γι' αυτό συνεχίζουμε να εξετάζουμε τα θέματα αυτά γιατί έχουμε ε, τέτοιες περιπτώσεις αλλά ε, δεν διερευνούμε μεμονωμένες περιπτώσεις και αυτό παραμένει η θέση μας. Okay. Floor to members, Mr. Τα μέλη. Ευχαριστώ. Άκουσα την αντίδραση της Κομισιόν και έχω μπερδευτεί. Δηλαδή έχουμε μία περίπτωση όπου λέει η Κομισιόν ότι εδώ η ελληνική κυβέρνηση δεν εφάρμοσε τους ευρωπαϊκούς νόμους. Για κάθε έργο, ακόμα και σε αυτό το τομέα, θα πρέπει να γίνεται εφαρμογή με βάση την νομοθεσία. Η Κομισιόν τι λέει. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα αν προκειμένου. Δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό το πράγμα και δεν το πιστεύω. Ξέρω περιπτώσεις συγκεκριμένες που είχαμε παρόμοια έργα και όπου υπήρχαν ε, παραβιάσεις και η Κομισιόν πρέπει να αναλάβει δράση εν προκειμένου και να κάνει κάτι. Γιατί εδώ έχουμε μια περίπτωση όπου ένα κράτος μέλος παραβιάζει την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία. Άρα χρειάζεται να, ληφθεί, ε, να αναλυφθεί η δράση. Γιατί από την έρευνα της Κομισιόν φαίνεται τι έγινε. Ακόμα και η παρουσίαση της αναφέρουσας το κατέδειξε αυτό. Λέω λοιπόν ότι πρέπει η αναφορά να παραμείνει ανοιχτή και όχι μόνο. Η Κομισιόν πρέπει να χρησιμοποιήσει κάθε μέτρο που είναι στη διάθεσή της για να φροντίσει αυτή η παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στο περιβαλλοντικό τομέα από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης να πάρει ένα τέλος. Κυρία Ούκεν. Συμφωνώ απόλυτα με τον προηγούμενο ομιλητή. Δεν θα έλεγα ότι σοκάρομαι, γιατί είναι κακή συνήθεια της Κομισιόν να κοιτάει το περιβαλλοντικό δίκαιο ως είναι κάτι που δεν πρέπει να το παίρνει κανείς στα σοβαρά στην Κομισιόν. Το έχουμε δει και ξαναδεί το έργο αυτό. Και σήμερα το πρωί ε, στην ετήσια έκθεση και, ε, λέμε και περάσαμε ένα ψήφισμα που λέει ότι αυτό πρέπει να σταματήσει. Η Κομισιόν πρέπει να καταλάβει ότι είναι θεματοφύλακα τη συνθήκη πρέπει να το δει πιο σοβαρά. Τι είναι αυτό να λέει αφήστε το στα εθνικά δικαστήρια. Άμα υπάρχει σαφής καταστρατήγηση του ενωσιακού δικαίου που περί αυτού πρόκειται εδώ. Ε, ή μπορεί να μην το ξέρουμε ακόμα, αλλά αν δεν καταπιαστείτε να το ερευνήσετε το θέμα... Και από ό,τι κατάλαβα, πρόκειται για ένα έργο ελληνικό που ερευνήθηκε. Αν προχωρήσουμε με έργα σε περιοχές Natura 2000, θα πρέπει να δικαιολογηθεί ότι δηλαδή είναι ε, πάρα πολύ, αναγκαίο, δεν γίνεται χωρίς αυτό και δεν υπάρχουν εναλλακτικά. Και στη Γερμανία ε, δείξατε την ίδια υπεροπτική στάση με τους νόμους του 2000, ότι δεν, είναι δικό σας θέμα. Natura 2000, ας πάει να ρυθμιστεί στο εθνικό επίπεδο, ε, δεν θα ασχοληθούμε εμείς. Όχι πρέπει να μείνει ανοιχτή η αναφορά και θα πρέπει να πάει στον Επίτροπο Σεύκοβιτς όταν θα έρθει την άλλη εβδομάδα. Είναι... Θα πρέπει να πείσουμε την Κομισιόν, να την πιέσουμε ότι είναι θεματοφύλακες της ε, συνθήκης. Δεν μπορεί να πλένουν τα χέρια τους σαν τον Πόντιο Πιλάτο και να μας στέλνουν όλους στα εθνικά δικαστήρια. Ε, να ένας από τους πολλούς λόγους που έχουν οι πολίτες για να δυσπιστούν απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Νικολάου Αλαβάνος. Ε, επαναλάβω κανένα από τα στοιχεία που έχουν δώσει οι προηγούμενοι ομιλητές, ούτε τα στοιχεία που έχει καταθέσει αναφέρουσα στην αναφορά της, τα οποία αξίζουν μελέτης ξανά. Ε, θέλω να πω όμως το εξή Είναι δεύτερη φορά στην Επιτροπή Αναφορών, μέσα σε ένα μήνα, όπου συζητούμε ένα ζήτημα ελληνικού ενδιαφέροντος, συγκεκριμένου θέματος, το οποίο έχει να κάνει με ε, βιομηχανική λειτουργία ή ε, εκμετάλλευση μέσα σε χώρο είτε προστατευόμενο από τα προγράμματα Natura, είτε χαρακτηρισμένο σαν ε, ιστορικής σημασίας, είτε ε, φυσικού κάλους Μιλάω για τις σκουριές που συζητήσαμε την προηγούμενη φορά και η απάντηση από την Κομισιόν είναι η ίδια πάνω κάτω ότι εν πάση περιπτώσει αρμόδιος είναι να λύσει τα ζητήματα η ελληνική νομοθεσία και ο Έλληνας ε, νομοθέτης και το δικαστικό σύστημα. Ε, είναι κατά την άποψή μας μια υποκριτική από μεριάς της Κομισιόν ε, τοποθέτηση καθώς όταν βάζει τα περιβαλλοντικά πλαίσια για παράδειγμα για τις ανανεώσιμες πηγές για το πώς θα γίνουν, ποιοι όμιλοι θα τα αξιοποιήσουν, ποιοι όμιλοι θα κάνουν τις επενδύσεις. Πληρώνει βαρύτατα ο ελληνικός λαός σε φορολογία, κλείνουν οι κρατικές επιχειρήσεις, πετιούνται χιλιάδες άνθρωποι στην ανεργία όπως γίνεται αυτή την περίοδο στη Δυτική Μακεδονία, πράγμα το οποίο είναι αποτέλεσμα της πολιτικής που εφαρμόσαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα να θυμίσω ότι είναι με νόμο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ που επιτρέπει την αλλαγή εύκολα της χρήσης γης για να γίνονται τέτοιου είδους επενδύσεις. Αλλά όταν διαμαρτύρονται οι πολίτες δικαίω για την περιβαλλοντική καταστροφή, για τις επιπτώσεις στην υγεία, τότε μνήπτει τα σχήρα τη. Εμείς σαν ΚΚΕ είμαστε αντίθετοι στην εγκατάσταση μονάδων ενεργειακής κάψης βιομάζας βιορευστών και σε αυτή την περιοχή, στο πλαίσιο του συνολικού αγώνα ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του ενεργειακού τομέα της χώρας μας, έχουμε αναδείξει το ζήτημα. Πέρυσι τέτοια εποχή καταθέσαμε ε, αναφορά στην Ελληνική Βουλή από Δημοτικό Συμβούλιο παρακείμενης περιοχής του Μεσολογγίου στο Ξηρόμερο για το ίδιο ζήτημα και θα συνεχίσουμε. Νομίζουμε ότι με τον τρόπο που γίνεται η ευρωενωσιακή νομοθεσία δεν μπορεί ούτε το περιβάλλον ούτε και τη ζωή και την υγεία των κατοίκων να προασπίσει γιατί όταν έχει να επιλέξει ανάμεσα στο, στα μεγάλα μονοπόλια που θέλει να ε, υπερασπιστεί και να σπρώξει στην κούρσα του ανταγωνισμού με άλλα τότε ανοίγει ο επικίνδυνο δρόμος με αυτές τις αρνητικές περιβαλλοντικές συνέπειε και πολλαπλέ δυσμενεί επιπτώσει για τους κατοίκους. Άρα κατά την άποψή μας νομίζουμε πρέπει να εξεταστούν τα στοιχεία που δίνονται, να μείνει ανοιχτή η αναφορά και να δούμε σε δεύτερο επίπεδο τι απαντήσει θα έχουμε. Γιατί, εν πάση περιπτώσει, λέγαμε το δίσεξα εξαμαρτίν ούκανδρο σοφού, αλλά το πολλάκι δεν ξέρω πού μα πηγαίνει. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Λαβάν Νικολάου και θα ήθελα και εγώ να πω δύο λόγια. Ε, πραγματικά είναι σοκαριστικό ε, που στην Κομισιόν ε, δεν αναφέρεται καθόλου στις επιπτώσεις που μπορεί να υπάρχουν και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε εθνικό επίπεδο. Είδαμε και από την αναφέρουσα πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα και πολλοί είναι οι συνάδελφοι οι οποίοι πραγματικά ε, ενδιαφέρονται για όλα τα περιβαλλοντικά ζητήματα και βάση φυσικά και του ενωσιακού δικαίου. Ε, ε μην λησμονούμε ότι έχουμε πλέον μπροστά μας ε, και το στρατηγικό σχεδιασμό αυτής της πράσινης συμφωνίας Green Deal. Βάσει των όσων ακούσαμε, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά και καλούμε την Κομισιόν να μελετήσει περαιτέρω τις καταγγελίες της αναφέρουσας και βεβαίως να δούμε κατά πόσον υπάρχει παραβίαση και του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και διεθνών συμβάσεων. Ξέχασα να σας ξαναδώσω το λόγο. Δύο λεπτάκια. Παρακαλούμε πάρα πολύ όμως να μην μιλάτε τόσο γρήγορα γιατί οι διερμηνείς δυσκολεύονται πάρα πολύ. Και ζητώ συγγνώμη από τους διερμηνείς, απλά είναι το πάθος. Έχω έρθει χθες από το Μεσολόγγι. Ε, θα ήθελα απλά να σχολιάσω ε, το, το θέμα που θίχθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η αδειοδότηση δόθηκε το 2014, δεν έγινε καμία διαβούλευση, δεν ζητήθηκε καμία γνώμη από την τοπική κοινωνία και τα εργοστάσια άρχισαν να κατασκευάζονται το 2017. Επομένως, η τοπική κοινωνία, αλλά και όποιος φορέας ήθελε να προβεί στον εθνικό δικαστή, έχασε τις προθεσμίες. Εμείς κάναμε ό,τι γινόταν στα εθνικά δικαστήρια, αλλά η απάντηση που παίρναμε δεν μπαίναν στην ουσία του ζητήματος, Μα ε, μας λόγω προθεσμίας. Γιατί, Γιατί δεν μας δόθηκε ποτέ ποτέ η δυνατότητα να το μάθουμε. Η έλλειψη αυτή διαβούλευση και το γεγονό ότι παραβιάζεται και το εθνικό αλλά και το ευρωπαϊκό δίκαιο στο κομμάτι αυτό, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό η τοπική κοινωνία να μαθαίνει το σχεδιασμό, να σχολιάζει και φυσικά είναι πολύ σημαντικό όταν υπάρχουν σχέδια όπως αυτά της ολοκληρωμένη χωρική επένδυσης να ακολουθούνται. Γιατί σε μια περιοχή που θέλει να στηρίξει τη γεωργία, την κτηνοτροφία, την αλληλεία και την ήπια οικοτουριστική ανάπτυξη δεν μπορείς μέσα στο εθνικό πάρκο το οποίο προστατεύεται από τόσε συνθήκε να πας να φτιάξει μονάδες που θα καίνε τη γανέλαια και χωρίς να έχεις κάνει και τις σωστές μελέτες. Επομένως, κατανοούμε ε, το σκεπτικό της Επιτροπής, παρόλα αυτά δεν μπορούμε με τίποτα να το στηρίξουμε ε, και από τη στιγμή που έχετε πάρει ήδη την απόφαση ε, για να παραμείνει ανοιχτή, αυτό θέλουμε κι εμεί και να πω ότι το Εθνικό Πάρκο ε, Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου Ετολικού ε, είναι το πλουσιότερο σε χλωρίδα και πανίδα ε, στην Ευρώπη. Εκεί βρίσκουν καταφύγιο πουλιά, εκεί υπάρχουν σπάνια φυτά και το να υπάρξουν και να δουλέψουν αυτές οι μονάδες υποβαθμίζουν καταρχήν την υγεία εμάς των πολιτών, κατά δεύτερον τις καλλιέργειες και κατά τρίτον τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής. Ευχαριστώ πολύ. Thank Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Δασκάλη. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι η πρότασή μας είναι να αφήσουμε ανοιχτή αυτή την αναφορά και καλούμε βεβαίως την Επιτροπή να διερευνήσει περαιτέρω αυτήν την αναφορά και την κατάσταση με τη δέουσα επιμέλεια και προσοχή. Ε, υπάρχει κάποια αντίρρηση. No, no, we, I'm sorry, we are running out. Ε, ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Δεν έχουμε χρόνο. Φαντάζομαι ότι ούτως ή άλλως θα σας πούν ποια είναι η απόφαση και νομίζω ότι θα ικανοποιηθείτε από την απόφασή μας. Άρα, άρα, ολοκληρώσαμε... Committee of Petitions and we switch to the coordinate. Και τώρα θα αρχίσει η συνεδρίαση των συντονιστών. So, Άρα, παρακαλώ να παραμείνουν στην αίθουσα μονάχα οι συντονιστές ή όσοι τους εκπροσωπούν. Όλοι οι υπόλοιποι παρακαλώ.